Συνάδελφοι, ας ε, ξεκινήσει η συνεδρίαση της Επιτροπής Μεταφορών. Έχετε το σχέδιο ημερήσιας διάταξης, να υποθέσω ότι είναι δεκτό. Αν ναι, ναι, σας ευχαριστώ. Μετά έχουμε την έγκριση των πρακτικών της 31ης Μαΐου και της 1ης Ιουνίου. Εγκρίνονται αυτά τα πρακτικά. Ευχαριστώ πολύ. Πριν περάσουμε στην έκθεση της κυρίας Γένσεν για τα ευφυή e e συστήματα μεταφορών, καλωσορίζω μια ομάδα Ολλανδών επισκεπτών από την ομάδα του κυρίου Βαντάλεν, προσκεκλημένη του κόμματος κυρίου Βαντάλεν. Καλώς ήρθατε. Είναι ενδιαφέρουσα η συζήτηση και ελπίζω κάτι να αποκομίσετε και πάντα χαιρόμαστε να έχουμε επισκέπτες στην Επιτροπή μας και καλεσμένους του κυρίου Φαντάλεν και ελπίζω να απολαύσετε τη συνεδρίασή μας. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Κυρία Γένσεν, ΕΦΗ, e συστήματα μεταφορών και θα εξετάσουμε τις τροπολογίες. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Γρήγορα πάμε. Γιατί δεν ε, έχουν κατατεθεί πολλές τροπολογίες και αυτές που κατατέθηκαν ε, δεν τις ε, συνιστώ. Υπάρχουν κάποιες τροπολογίες, δύο πρώτα από τους Γάλλους συναδέλφους που αντικατοτρίζουν κάποιους, κάποιες γαλλικές ανησυχίες. αλλά βεβαίω το σύστημα το γαλλικό δεν θα είναι διαλειτουργικό με τα νέα συστήματα. Και αντιλαμβάνομαι την αγωνία του κυρίου και, και ότι μπορεί να τις αποσύρει. Γιατί η ενισχύα του ήταν το ότι αυτά τα οποία, στα οποία έχει επενδύσει η Γαλλία θα μπορούν να συνδεθούν με το νέο σύστημα. αλλά νομίζω πως η Κομισιόν εγγυάται πως δεν θα υπάρχει πρόβλημα για τη Γαλλία. Οπότε με δεδομένο αυτό ελπίζω αύριο να μπορέσουμε να ψηφίσουμε χωρίς ίσως τις δύο αυτές τροπολογίες. Θα απαντήσει ο κ. Εγώ προτείνω να ψηφίσουμε όχι στις δύο τροπολογίες. Αυτή είναι η σύστασή μου. Και μετά θα μπορέσουμε να ρυθμίσουμε αυτό το, το ζήτημα και να περάσουμε στο πώς θα έχουμε πιο ευφυή συστήματα μεταφορών. Ευχαριστώ κυρία Τικάου. Uh, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας uh, ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ με τα όσα είπε η κυρία Γένσεν. Όντω, εργαστήκαμε πάρα πολύ προκειμένου να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε αυτή τη συμβαστική πρόταση και πιστεύω ότι θα πρέπει να καταψηφίσουμε τις δύο τροπολογίες στις οποίες αναφέρθηκε η κυρία Γένσεν. Το καλύτερο βέβαια θα ήταν να αποσύρονταν οι τροπολογίες αυτές. Πιστεύω ότι μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να εγκρίνουμε αυτή τη δέσμη μέτρων η οποία είναι απαραίτητη. Ευχαριστώ. Thank Καφέ θέλετε πρώτα, πρωτού μιλήσετε, γιατί άμα φύγουνε φύγανε, δεν θα ξανάρθουνε ή τώρα ποτέ λοιπόν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αποσύρω τις τροπολογίες μου. Τροπολογίες που είχαν ακριβώς αυτό το στόχο που περιέγραψε η Άννα. Υπήρχε μια φυσιμία την οποία είχε εντοπίσει προφορικά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί ε, τα, αυτά τα ευφύ συστήματα μεταφορών θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη από την εθνική νομοθεσία και δεν θα ήταν ένα σύστημα το οποίο θα επιβελόταν απλώς εκ των άνω. Αποσύρω πάντως τροπολογίες μου κύριε Πρόεδρε όπως ζήτησε άλλωστε και η συγγήτρια. Ευχαριστώ. Thank you very much, Dominic. Ευχαριστώ, Ντομινίκ. Από την Κομισιόν ο κύριος Πακέ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, μπορώ να επιβεβαιώσω πως ε, τα υπάρχοντα συστήματα θα ενσωματωθούν πλήρως στο σύστημα Equal που θα δημιουργηθεί και ζητώ συγγνώμη αν υπήρχε αμφισημία, αλλά δεν νομίζω πως υπάρχει λόγος ανησυχίας. Σας ευχαριστώ. Κυρία Γένσεν, θέλετε να δευτερολογήσετε. Όχι, νομίζω πως όλα ακούστηκαν. Ευχαριστούμε, Ντομινίκ, που αποσύρεις ε, τις ε, τροπολογίες σου. Έτσι γίνονται απλούστερα τα πράγματα για αύριο. Και μετά θα έχουμε την ψηφοφορία στην Ολομέλεια τον Ιούλιο. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενο σημείο είναι η δική μου έκθεση στατιστικές καταγραφές για τις θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών. Εξέταση τροπολογιών. Θα θυμάστε πως αυτή είναι μία από αυτές τις εκθέσεις που με μεγάλη γενεοδορία που και που δίνεται στον πρόεδρο όταν δεν θέλει κανείς άλλος να κάνει καμία έκθεση, οπότε προσπάθησα να ετοιμάσω μία έκθεση. Η οδηγία η οποία τροποποιείται αφορά έναν κανονισμό που ισχύει ήδη για τις θαλάσσιες και ποτάμιες μεταφορές το άρθρο 2α που καλύπτει εν μέρη μόνο τις θαλάσσιες μεταφορές και τονίζω εδώ το θαλάσσιες στο πλαίσιο αυτό πρέπει να επισημάνουμε πως η Κομισιόν είναι υποχρεωμένη να καταπτύσσει ένα κατάλογο λιμένων εφαρμογής αυτής της οδηγίας. Επειδή η απόφαση αυτή λαμβάνεται σύμφωνα με τη διαδικασία της ε, συναπόφασης, θα ενισχυθεί η συμμετοχή του Κοινοβουλίου για τον κατάλογο αυτών των λιμένων, εάν οι τροπολογίες αυτές στο, ε, σύμφωνα με τις πράξεις κατεξιοδότηση υιοθετηθούν. Υπήρχαν ε, κάποια πράγματα καθώς έλεγαν πως ε, θα είναι ένα επιπλέον διοικητικό βάρος συλλογής στατιστικών δεδομένων, αλλά ούτως ή άλλως σε μεγάλο βαθμό συλλέγονται αυτές τις πληροφορίες από τις Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες. Οπότε δεν νομίζω να υπάρχει κανένα πρόβλημα στο να ε, μιλάμε για περαιτέρω διοικητικό βάρος, αυτή η δουλειά ήδη γίνεται. Υπήρχε μια τροπολογία που κατέθεσε η κυρία Τικαού και είναι κάτι που καλύπτεται νομίζω όπως έχω καταλάβει και η κυρία Τικαού ευγενικότατα δέχτηκε να αποσύρει την τροπολογία της. Οι τροπολογίες για τις πράξεις κάτω εξουσιοδότηση, εάν υιοθετηθούν, οι δικές μου δηλαδή τροπολογίες, θα δώσουν στο Κοινοβούλιο μεγαλύτερο λόγο για να αποφασίζει ποιοι λιμένες θα συμπεριληφθούν στον κατάλογο. Επειδή αυτή η απόφαση λαμβάνεται σύμφωνα με τη διαδικασία της επιτροπολογίας, σας ζητάω να υποστηρίξετε αυτές τις τροπολογίες για να ενισχυθεί η θέση του Κοινοβουλίου σε σχέση με την... τις πράξεις αυτές κατά εξουσιοδότηση, όπως θα τις λέμε από εδώ και μπρος. Οπότε, ε, θα μείνουμε σε αυτά. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Ο κύριο Κούν, η κυρία Τικάου και ο κύριος Μάης έχουν ζητήσει το λόγο. Κύριε Κούν, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την δουλειά που έχετε κάνει εδώ πέρα, γιατί είναι αναγκαίο να γίνεται αυτή η κοινή συλλογή στατιστικών δεδομένων για τις μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών εντός της Ένωσης. Είναι βασική προϋπόθεση για να είναι αποτελεσματική η διατροπική μεταφορά, δηλαδή εκεί όπου υπάρχει μεταφορά μου πολλά μέσα, να ξέρουμε ποιες είναι οι ροές οι εμπορευματικές στην Ευρώπη και να γίνουν οι απαραίτητες προβλέψεις για τους ε, σιδηρόδρομους και να δούμε τι θα συνδεθεί στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε μια βάση με δεδομένα. Γι' αυτό γίνεται με αυτή την οδηγία. 18 κράτη-μέλη συλλέγουν ήδη αυτά τα δεδομένα. Θέλουμε λοιπόν όλα τα κράτη τα οποία αφορά αυτή η οδηγία να συλλέγουν αυτά τα δεδομένα πλην ε, πέντε κρατών βεβαίως που δεν έχουν πρόσβαση στη θάλασσα οπότε δεν γίνεται λόγος περιλημμένων. Θεωρώ πολύ θετικό και ευχαριστώ τον εισηγητή για το ότι αυτά τα οποία είναι απαραίτητα από πλευράς ε, επιτροπολογίας να καλύπτονται με τροπολογίες έτσι ώστε να έχουμε την ε, θέση, την δυνατότητα να ανακτήσουμε την ομοθετική ισχύ που έχει πάρει η Κομισιόν. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικές οι τροπολογίες και συμφωνούμε με αυτές και ευχαριστούμε και την κυρία Τικάου που τις απέσυρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Τικάου. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Μου είπατε ότι καλύπτεται η τροπολογία μου ήδη από το κείμενο, κύριε Πρόεδρε, και συγγητά, επομένως μπορώ να αποσύρω την τροπολογία μου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μάισνερ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Συχνά ο Πρόεδρος έχει αυτές τις εκθέσεις που δεν είναι και οι πιο συναρπαστικές, αλλά βεβαίως δεν σημαίνει πως δεν είναι σημαντικές. Είναι σημαντικές γιατί πρέπει να έχουμε δεδομένα. Αλλά νομίζω πως ο κύριος Σίμψον το είπε αναλυτικά γιατί θέλει να κάνει αυτές τις ε, τροπολογίες για να ενισχύσει και τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου. Το έχει επιτύχει αυτό, γι' αυτό δεν έχουμε καμία τροπολογία και είμαστε ε, βεβαίως ικανοποιημένοι με τον Πρόεδρο, τουλάχιστον όσον αφορά αυτή την έκθεση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, είστε τόσο ευγενικοί. Κυρία Λίχτεμπέργκερ, ευχαριστώ. Εγώ βεβαίως επειδή προέρχομαι από ένα περίκλειστο κράτος δεν θα πω πάρα πολλά. Απλά ένα πράγμα που ξέρω από τα σχετικά στατιστικά στοιχεία είναι το ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη υστέρηση. Δηλαδή έχουμε δεδομένα του 2005-2006. Δεν ξέρω αν μπορούμε να επιταχύνουμε λίγο τη συλλογή και δεύτερον είμαι πεπισμένη πως ακριβώς λόγω της επιτροπολογίας θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την ποιότητα των δεδομένων και με την ταχύτητα των δεδομένων. Γιατί το να κοιτάμε παλαιότερα έτη δεν έχει νόημα. Μιλάμε έτσι για στατιστικά στοιχεία που αναφέρονται σε παλαιότερα έτη πρώτης οικονομικής κρίσης και δεν έχουν πλέον κανένα νόημα. Εντάξει, ευχαριστώ σωστό αυτό που είπατε. Για να επιταχύνουμε τη διαδικασία. Πολύ σωστό. Ακριβώς επειδή είναι επιτροπολογία. Για την Επιτροπή κύριος Μούρο. Ναι, ναι, σας βλέπω. Thank you, Mr. Chairman. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρο, Πρόεδρε. Αμερίνη ονομάζομαι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί με τις 8 αυτές τροπολογίες. Χαίρεται επίσης που η ενάτη τροπολογία έχει αποσυρθεί. Και όσον αφορά τα δεδομένα, μπορώ να σας πω ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα και το 2009. Θα δημοσιεύσουμε αυτά τα πρώτα αποτελέσματα. Επομένω μπορούμε να σας δώσουμε και πιο πρόσφατα δεδομένα όπως ζητήσατε. Πρόεδρος, Είδατε, δύο φράσεις είπατε και τα πάντα επιταχύνονται, τα πάντα λύνονται. Σας ευχαριστούμε πολύ. Το χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής. Αύριο θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή και στη συνέχεια θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου. Πολύ ωραία, συμφωνούμε όλοι. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, το εκτιμώ ιδιαιτέρως και περνάμε στη συνέχεια στον καθορισμό προτύπων για τις επιδόσεις των καινούριων ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων όσον αφορά τις εκπομπές. Εισηγητής είναι ο κύριος Βλάσακ. Θα θυμάστε ότι δεν μπορούσαμε να συζητήσουμε τη γνωμοδότησή σας την προηγούμενη φορά γιατί ήσταν απόν. Έχετε τώρα το λόγο κύριε Βλάσακ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να, πω και εγώ κάποια λόγια για το σημαντικό αυτό ζήτημα. Ζήτημα το οποίο οδήγησε σε πάρα πολλές ε, συζητήσεις και σε πάρα πολλές προτάσεις. Προσπάθησα να παρουσιάσω περισσότερο τη σκοπιά της Επιτροπής Μεταφορών στη γνωμοδότηση αυτή, θέτας κατά μέρος τα περιβαλλοντικά ζητήματα, εφόσον με αυτά ασχολείται η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Θέλησα εγώ να κάνω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λίγο πιο λογική όσον αφορά την υφιστάμενη οικονομική κρίση και όσον αφορά τις δυνατότητες της αυτοκινητοβιομηχανίας. Βασίστηκα σε κάποιες συζητήσεις που είχαμε με πολλούς συναδέλφους, καθώς επίσης και με διάφορα ερευνητικά κέντρα και στις συζητήσεις αυτές Μίλησα και με τους κοιόδης συγητές, τους οποίους θα ήθελα να ευχαριστήσω. Τον κύριο Ρικέ, τον κύριο Παζόν, τον κύριο Στέρξ, τον κύριο Κάμερον και την κυρία Βίλς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν για την πολύ καλή του συνεργασία. Νομίζω ότι θα πρέπει ακριβώς αυτή την προσέγγιση να ακολουθούμε κάθε φορά που καλούμεθα να συζητήσουμε για ένα συγκεκριμένο ζήτημα, ακόμα και αν δεν συμφωνούμε εξ αρχής. Κατά την άποψή μας, επιθυμούσαμε να είχαμε μια προσέγγιση πιο ορθολογική, πιο λογική, ενώ οι υπόλοιποι συνάδελφοι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλουν να προχωρήσουν πιο φιλόδοξα. Θα δείτε ότι υπάρχουν διάφορες συμβαστικές τροπολογίες που αντικατοπτρίζουν και τη συνένεση που έχουμε πετύχει και ελπίζω θα καταφέρετε να στηρίξετε τις τροπολογίες αυτές. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να εγκρίνουμε τη γνωμοδότηση αυτή έτσι ώστε να καταφέρουμε να στείλουμε ένα σαφές, ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Λοιπόν, ποιες είναι αυτές οι συμβαστικές τροπολογίες οι οποίες σας προτείνουμε. Η πρώτη έχει να κάνει με το όριο των 175 γραμμαρίων διοξιδίου του άνθρακα ένα χιλιόμετρο. Το στόχο αυτόν. Εμείς θα θέλαμε να μεταθέσουμε την προθεσμία μέχρι το 2014 και θα θέλαμε να έχουμε ένα μηχανισμό λίγο πιο ευέλικτο όσον αφορά τις κυρώσεις για την παραβίαση του στόχου αυτού. Η δεύτερη συμβαστική τροπολογία έχει να κάνει με το στόχο των 135 γραμμαρίων διοξιδίου του άνθρακα ένα χιλιόμετρο. Θεωρούμε ότι ο στόχος αυτός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει από το 2022 και μετά. Η τρίτη συμβαστική τροπολογία που έχουμε προτείνει είναι μείωση των προστήμων από 120 ευρώ σε 95 ευρώ. Κατά αυτόν τον τρόπο ευθυγραμμιζόμαστε με την οδηγία που έχει να κάνει με τα επιβατηγά οχήματα. Δεν νομίζω ότι σε καμία περίπτωση θα πρέπει να δημιουργούμε ένα σύστημα το οποίο θα εισάγει διακριτική μεταχείριση μεταξύ των οχημάτων. Η τέταρτη συμβαστική τροπολογία έχει να κάνει με τη χρήση των εσόδων από τα πρόστιμα και πώς τα έσοδα αυτά θα πρέπει να επενδύονται σε νέες τεχνολογίες, έτσι ώστε να καταφέρουμε μέσω των νέων αυτών τεχνολογιών να μειώσουμε τον αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον. Η τελευταία συμβαστική τροπολογία, η ε, είναι αυτή η οποία δεν χαίρει πλήρους υποστήριξης από όλες τις πολιτικές ομάδες και έχει να κάνει με τα όρια ταχύτητας ή τον περιορισμό της ταχύτητας αν θέλετε. Ακολουθώντας τον κανονισμό SMART πιστεύω ότι ε, θα πρέπει να έχουμε περιορισμό της ταχύτητας μόνο αφού γίνει μια αξιολόγηση αντικτύπου η οποία θα πρέπει να γίνει μόνο όταν τροποποιηθεί ο κανονισμός 92 κάθετο, κάθετος 6 που μιλάει για περιορισμό της ταχύτητας, για όρια ταχύτητας. Αυτές λοιπόν οι συμβαστικές μας τροπολογίες, οι συμβαστικές μας προτάσεις και σας προτείνω να γίνει μια ψηφοφορία on για τις ε, τροπολογίες αυτές και να μην δημιουργήσουμε ξεχωριστές τροπολογίες, να μην, να μην κάνουμε ξεχωριστή ψηφοφορία για τις τροπολογίες αυτές, γιατί θεωρώ ότι αυτό θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, σκιώδεις ηγητές για άλλη μια φορά που με εμπιστεύτηκαν που μου δώσαν τη δυνατότητα να συντάξω την γνωμοδότηση αυτή και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Μάθιου Μπράουν από την Γραμματεία για την ανακοίνωση που έκανε. Θα ήθελα επίσης να πω για μία ακόμη φορά ότι ε, στόχος μας είναι να καταλήξουμε σε κάποιες συμβαστικές προτάσεις. Αυτό ακριβώς έχετε μπροστά σας αυτή τη στιγμή και δεν ε, συμφωνώ απαραίτητα απόλυτα με όλες αυτές τις συμβαστικές προτάσεις. Σε ορισμένα σημεία θα απέχω λοιπόν από την ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ κύριε Βλάσακ. Κατόπιν έχουμε τον κύριο Ρίκε για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ τον κύριο Φλάσακ, κύριε Πρόεδρε, και για την εργασία του και τη διάθεση που έδειξε για συμβαστικές λύσεις, γιατί δέχτηκε και συμβαστικές λύσεις που δεν του άρεσαν ενδεχόμενα και τόσο έτσι, μέσες. Αυτό βοήθησε για την επιτυχία όλων αυτών εδώ και είναι μια σημαντική απόφαση γιατί έχει να κάνει και με το περιβάλλον και με τη βιομηχανία. Και είτε θα έχουμε μια πτυχή του περιβάλλοντος εντάξει σχετικά με την ε, εκπομπή παρομοίων αερίων ε, πάνω σε αυτό και μόνο και κάτι ιδιαίτερα δεσμευτικό για αυτές τις εκπομπές ε, που θα είναι εις βάρος βέβαια της μηχανίας είτε θα δούμε τα πράγματα από οικονομικής πλευράς και θα προσπαθήσουμε να μην πιέσουμε τόσο την βιομηχανία και ε, το θέμα των τομέα των αυτοκίνητων Είχαμε 70, 170 τροπολογίες, διάφορες, πολλές, ε, ήταν από την πιο οικονομική μέχρι την πιο οικολογική, έτσι, ακόμα και μέσω όλων των πολιτικών ομάδων ε, και είναι, υπήρχε ένας μεγάλος κίνδυνος να μην ψηφιστεί καμία τροπολογία γιατί δεν θα ε, συγκέντρωνε πλειοψηφία, θα ήταν κάτι το καταστροφικό, δεν θα μπορούσαμε να γνωμοδοτήσουμε έτσι, ενώ η γνωμοδότησή μας πάνω σε αυτό το θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντική, είτε θα ερχόταν όλοι και θα νέρωναν το κρασί τους κάπως όπως λέμε και θα επέβαλαν τροπολογίες που βέβαια δεν θα ήταν ικανοποιητικέ πλήρως για όλους αλλά θα αποτελούσαν σε μέσα συμβιβαστικές λύσεις και για μας μια σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων ε, σε σχέση με το περιβάλλον πάντα και ακόμα μια κάποια υποχρέωση να μπορούν να είναι ανταγωνιστική η βιομηχανία και στα πλαίσια αυτής της κρίσης να μην δημιουργούσε ιδιαίτερες δυσκολίες ε, στην ε, οικονομία μας. Αυτά και ολοκληρώνοντας η ομάδα μου όλες αυτές οι συμβαστικές λύσεις που προτάθηκαν τις υποστηρίζει. Βέβαια θα έχουμε και διάφορες άλλες τροπολογίες που θα μπορούσαν να διευκρινίσουν τα πράγματα σε διάφορες πτυχές της έκθεσης και που ίσως μέσω και ξεχωριστής ψηφοφορίας αλλά οι συμβαστικές λύσεις ελπίζω ότι θα συγκεντρώσουν ιδιαίτερη πλειοψηφία, ευρεία πλειοψηφία για να είναι κάτι το ισορροπημένο και να μπορεί να γίνει ε, δεκτό από τους συναδέλφους μας της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Φαγιόν για τους σοσιαλδημοκράτες. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον εισηγητή τον κύριο Βλάσα και τους κοιόδης εισηγητές. Θα ήθελα να πω πως η γνωμοδότηση αυτή βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντική και αποδείχτηκε αυτό ότι τις τελευταίες εβδομάδες όλοι είχαν πολλές συζητήσεις με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και έπρεπε να καταλήξουμε σε πολύ σημαντικές συμβαστικές λύσεις για να έχουμε αύριο μια καλή ψηφοφορία για την ομάδα μας και για εμένα προσωπικά νομίζω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να παραμείνουμε φιλόδοξοι στο μακροπρόθεσμο στόχο μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Για μένα δύο πράγματα είναι σημαντικά. Η κίνηση αυτών των οχημάτων αυξάνεται, των ελαφρών εμπορικών οχημάτων και η ε, εκπομπές αυτές αυξάνονται όσον αφορά αυτά τα οχήματα με τον υψηλότερο ρυθμό Οπότε πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι και βέβαια ως συμβαστική λύση προτείνει ο εισηγητής είναι να καθυστερήσουμε κατά δύο χρόνια τα 135 γραμμάρια ε, να πάει στο 2022. Νομίζω είναι ήδη τεράστια παραχώρηση αυτή, αλλά στην Επιτροπή Μεταφορών εμείς είμαστε αυτοί που θα κάνουμε την πρώτη ψηφοφορία και οι άλλες επιτροπές θα ακολουθήσουν. Οπότε πρέπει να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Οπότε χαίρομαι για το ότι τουλάχιστον προσπαθούμε να παραμείνουμε παρά τα όσα μας είπε η αυτοκίνητο μηχανία. Καταφέραμε να επιτύχουμε αυτό τον συμβιβασμό και από την άλλη Έχουμε τον ενδιάμεσο στόχο, τα 175 με διαφορετική ε, εφαρμογή. Νομίζω είναι ένας καλός συμβασμός. Κάτι άλλο που θα ήθελα να θίξω. Εγώ και η ομάδα μου θα θέλαμε να μείνουμε στα 120 ευρώ για το πρόστιμο και αυτό βεβαίως αφορά το οριακό κόστος συμμόρφωσης που μιλάμε δηλαδή για 120 αναγραμμάριο ανά χιλιόμετρο. Και βεβαίως το ζήτημα της ταχύτητας το οποίο αναφέρθηκε γνωρίζω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό Διαβάζουμε πολλά στατιστικά στοιχεία. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό είναι το ιδανικότερο που μπορούμε να κάνουμε, αλλά το να μειωθεί η ταχύτητα, ακόμα και στα ελαφρά οχήματα, από τη μία βεβαίως μπορεί να μειώσει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, από την άλλη όταν συζητάμε την ασφάλεια στους δρόμους μας είναι εξίσου σημαντικό. Οπότε θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την συνεργασία και εγώ προσωπικά θα ήθελα να δω ένα θετικό αποτέλεσμα. Και υπάρχει ο και ενισχύει για το περιβάλλον και θα θέλαμε να δούμε πως ακόμα και η αυτοκίνητο που αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα να δείξει ότι παίζει και αυτή ένα σημαντικό ρόλο στη μείωση των εκπομπών στο περιβάλλον μας. Ευχαριστώ. Um, Ευχαριστούμε κυρία Φαγιόν. Ο κύριος Στέρξ για τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ευχαριστήσω την κυρία Βλάσακ για τη δουλειά που έκανε μίλησε πάρα πολύ με τους ε, συναδέλφους, ε, είχαμε ανταλλάξει ιδέες, ε, συγκρίναμε τα πράγματα και νομίζω πως πολλές από τις συμβαστικές αυτές λύσεις μπορούμε να τις στηρίξουμε. Και η πρόταση της Κομισιόν έρχεται την κατάλληλη στιγμή μετά από τα όσα έγιναν για τα επιβατικά οχήματα πρέπει να κάνουμε και κάτι για τα επαγγελματικά και είναι κάτι το σημαντικό αυτό. Πρέπει να φροντίσουμε ε, να μειωθούν οι εκπομπές. Την ε, Α νομίζω μπορούμε να την συμφωνήσουμε για τα 175 από το 2017 και μετά. Τώρα, πρέπει να παραμείνει νομίζω ο στόχος που υπάρχει στην συμβαστική λύση. Μίλησα πάρα πολύ με τους κατασκευαστές και είδα πως εργάζονται με, δεκαετούς, με δεκαετής κύκλους και ο επόμενος κύκλος θα ξεκινήσει σε κάνα δύο χρόνια. Οπότε το 2020 δεν είναι παράλογο, αλλά πρέπει να υπάρξει εκεί πέρα μια πραγματική μείωση και να παραμείνουμε κάτω από τα 135 γραμμάρια. Επίσης για το πού πρέπει να πάνε τα έσοδα από τα πρόστιμα. Δεν συμφωνούμε με το να μειωθούν τα πρόστιμα. Δεν θέλουμε να πάνε στο ίδιο επίπεδο με αυτά των αυτοκινήτων. Θεωρώ πως σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να παραμείνει η πρόταση της Κομισιόν. Όσον αφορά δε τον περιορισμό της ταχύτητας, δεν είναι καλή ιδέα ε, το να γίνει κάτι το εθελοντικό, γιατί σε ένα κράτος μέλος θα έχουμε διαφορετικό όχημα από ότι σε ένα άλλο κράτος μέλος. Νομίζω καλύτερο είναι, μου φαίνεται, και είναι και πρακτικό για την εσωτερική αγορά και τους κατασκευαστές, να έχουμε μία αγορά. Ή έχουμε δηλαδή όριο ή δεν έχουμε. Και πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Το εύκολο είναι να πούμε κάντε ό,τι θέλετε. Αλλά το να ισχύει κάτι σε μια χώρα και όχι σε μια άλλη δεν είναι σωστό. Είμαι υπόρ της τροπολογίας λοιπόν της κυρίας Φερχόνεν και Σαΐντ Ελχαντραουή. Νομίζω ότι είναι υπαριθμόν 100. Αλλά νομίζω είναι κάτω από τα 100 ε, σε αυτό είμαι υπέρ και όχι υπέρ της συμβαστικής λύσης. Επίσης είμαι υπέρ της πρότασης του εισηγητού για τα οχήματα πολλαπλών ε, φάσεων. Επίσης δεν ξέρω αν συμφωνώ με τη δυνατότητα να, κάνουν, να μοιραστούν κάποια πράγματα. Ε, και εννοώ εδώ πέρα βεβαίω τα επιβατικά και τα φορτηγά οι κατασκευαστές. Όχι, πρέπει να υπάρχει ε, διάσπαση ανακατηγορία για να υπάρχει και τίμιος ανταγωνισμός μεταξύ αυτών που φτιάχνουν και που δεν φτιάχνουν φορτηγά. Επίσης, ε, να πω πως θα πρέπει να έχουμε μια ξεκάθαρη θέση ως Επιτροπή Μεταφορών, γιατί αν δούμε το τι γίνεται και ε, σε σχέση με το περιβάλλον, αλλά και να δείξουμε ότι είμαστε ρεαλιστές για το μέλλον της βιομηχανίας. Να τους ξεκαθαρίσουμε δηλαδή ότι τους ακούσαμε μέσω της επιμήγυνσης των ορίων και η Επιτροπή Περιβάλλοντος και πιθανώς η Ολομέλεια θα α, ε, μας ακολουθήσει. Αλλά νομίζω πως αυτό το οποίο ρώτησε ε, και ζήτησε α, ε, μέσα στην Κομισιόν πηγαίνει πολύ παραπέρα από το που έχουμε πάει εμείς μέχρι στιγμής και νομίζω μπορούμε να πούμε άρα πως δεν είναι πολύ φιλόδοξος αυτός ο στόχος. Δηλαδή τηρούμε το 135 γραμμάρια και πάμε δύο χρόνια παραπέρα. Νομίζω είναι ένας ρεαλιστικός συμβασμός. Ευχαριστώ. Κύριε Dank. Äh, Ευχαριστώ. Όπως φαντάζεστε δεν συμφωνώ με τον συμβασμό, δεν κάλεσε καν τους πράσινους ε, ο εισηγητής. Ε, έφερε αυτούς που ήθελαν να καθυστερήσουν και αυτούς που ήθελαν να καθυστερήσουν πάρα πολύ την ε, διαδικασία. Οπότε δεν μπορώ να συμφωνήσω με κανένα από αυτούς τους στόχους. Όλος ο φάκελος δυστυχώς είναι μία από αυτές τις αποδείξεις ε, για το ότι η Επιτροπή μας ε, δεν είναι ρεαλιστική αλλά φρενάρει τα πράγματα στο περιβάλλον γιατί οι νέες μελέτες αποδεικνύουν πως ε, τα 135 θα μπορούσαν να έχουν επιτευχθεί τα 175 πρώτα απ' όλα εάν γίνει πρώτα απ' όλα μία ομοίωση τους μεγέθους. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός ε, όσον αφορά τις δυνατότητες αυτών των ελαφρών φορτηγών που είναι καταστροφική και δεν φέρνει τίποτα. Επίσης, εάν μας λέτε να γίνει και αντί, μελέτη αντικτύπου για τη μείωση της ταχύτητας γίνονται παράλογα τα πράγματα. Γιατί το τι ε, σημαίνει χαμηλότερη ταχύτητα, αυτό το ξέρουμε είναι γνωστό. Έχει θετικές επιπτώσεις στην ασφάλεια, στο περιβάλλον, αν υπάρχουν όρια ταχύτητας και ειδικά με αυτή την κατηγορία οχημάτων δυστυχώς διαπιστώνουμε πως είναι πάρα πολύ πιεσμένα, γίνουν αυτές οι γρήγορες μεταφορές, αγνοούν τα όρια ταχύτητας, αγνοούν ε, το χρόνο ανάπαυσης, ευνοούνται στα διόδια, γι' αυτό και αυξάνεται αυτός ο κλάδος των αυτοκινήτων και εμείς, εσείς, θέλετε να ζώσετε άλλα δύο χρόνια. Τεχνικά είναι ξεκάθαρο, γίνονται αυτά τα πράγματα ήδη και αν η αυτοκινητοβιομηχανία έρχεται και μας λέει πως δεν είναι, είναι απλό το, το τι γίνεται. Είναι προς το συμφέρον τους να το καθυστερήσουν, γιατί η καινοτομία κοστίζει. το εάν θα χάσουν και σε ανταγωνιστικότητα είναι ένα γεγονός που δεν πρέπει να αγνοήσουμε. Οπότε είμαι πολύ απογοητευμένη από αυτή την έκθεση και ε, δεν μπορώ να ταυτιστώ εγώ με αυτή τη συμβαστική λύση. Το pooling, δε, το να βάζουμε όλα τα μάξια μαζί που είναι η μεγάλη δικαιολογία της αυτοκινητοβιομηχανίας και θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερες αναβολές της ε, αποτελεσματικότητας των οχημάτων όσον αφορά το περιβάλλον ε, είναι σαφές. Οπότε το θεωρώ λάθος να ευνοείται μια κατηγορία οχημάτων έτσι, γιατί αυτό κάνουμε εδώ πέρα και εκεί πέρα ο ανταγωνισμός ε, μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών φορτηγών εντείνεται και δεν θα επιτύχουμε τίποτα για το περιβάλλον. Και αν αυτό το τίποτα το επιτύχουμε και ακόμα αργότερα, δεν ε, ωφελούμε το περιβάλλον. Κάνουμε ένα βήμα πίσω από το εφικτό και έχουμε ήδη την εμπειρία πως δεν αντιδρά από μόνο τη η αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά μόνο, μόνο μετά από πίεση. Και τότε όμως πολύ αποτελεσματικά και έτσι είναι πιο ανταγωνιστικά τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα. Θεωρώ λοιπόν πως εδώ πέρα αυτός ο δρόμος που ακολουθούμε είναι λάθος, δεν θα τον ακολουθήσουμε και θα δούμε τώρα με την ταχύτητα τι θα γίνει με τις προφορικές τροπολογίες γιατί δεν ξέρω Εάν δείτε τι γίνεται στους αυτοκινητόδρομους και σας περνάνε έτσι αυτοί οι επικίνδυνοι τύποι, τι να σας πω, εγώ σας εύχομαι καλή τύχη για την οδική ασφάλεια. Απλά να ξέρετε τι έχετε κάνει. Ευχαριστώ, κύριο Αλχαντραούλη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος γιατί οι συνάδελφοι είπαν αρκετά. Συμφωνώ με το ότι είναι σημαντικό το ότι επιτύχαμε κάποιες συμβαστικές λύσεις γιατί αλλιώς δεν θα είχαμε μια κοινή θέση. Βεβαίως πρέπει να δούμε τον χρόνο όταν θα ισχύσουν αυτές οι ε, εκπομπές ως, ε, όπως δε και ο κύριος Στέρξ ε, δεν είμαι υπέρ του να χαμηλώσουν τα, τα πρόστιμα. Νομίζω η Κομισιόν εδώ πέρα έχει κάνει μία σειρά καλών προτάσεων στις οποίες θα πρέπει να μείνουμε και τέλος να επανέλθω στον περιορισμό ταχύτητας. Δεν θα είναι καλό να το κάνουμε αυτό εθελοντικά. Το ανέφερε νομίζω ο συνάδελφος. Ε, να σου πω την αλήθεια, αυτό είναι κάτι που πρέπει να το ρυθμίσουμε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, να μην το αφήσουμε σε κάποια κράτη-μέλη μόνο. Γιατί έτσι δεν, δεν θα αλλάξει τίποτα. Εδώ πέρα μιλάμε για μια τεχνική ρύθμιση που θα πρέπει ε, να καταστήσει τεχνικά δύνατο να πάει κανείς πολύ γρήγορα. Και υπάρχει και εδώ πέρα η περιβαλλοντική πτυχή. Υπάρχουν μελέτες που αποδεικνύουν πως οι εκπομπές θα μειωθούν έτσι. Αλλά είναι και ζήτημα οδικής ασφάλειας. Όταν γκαζώνουν ε, τα αυτοκίνητα και όταν έχουν πάρα πολύ μεγάλη ισχύ, Εντάξει, μπορούν να μεταφέρουν και περισσότερα πράγματα, αλλά δεν μεταφέρουν περισσότερα πράγματα. Συνήθω πάνε απλά πιο γρήγορα. Οπότε θα πρέπει να δούμε τεχνικά ποιοι είναι οι, οι κανόνες. Ε, γνωρίζετε και τι γίνεται και μετά των 12 τόνων. Εκεί πέρα υπάρχει περιορισμός. Νομίζω θα πρέπει να μπορέσουμε αύριο να στείλουμε ως Επιτροπή ένα σαφές μήνυμα στους υπόλοιπους ε, συναδέλφους μας. Ευχαριστώ κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα είμαι σύντομη. Ο Ντίρκ Στέρξ νομίζω τοποθετήθηκε για τους φιλελεύθερους και τον υποστηρίζω απολύτως. Ήταν δύσκολο εδώ πέρα να βρούμε μια σωστή ισορροπία μεταξύ προστασίας του περιβάλλοντος, την οποία βέβαια θέλουμε να επιτύχουμε. Γνωρίζουμε πως ε, εκεί πέρα έχει μεγάλη συνεισφορά η αυτοκίνητο μηχανία και να δούμε και πώς θα αντιδράσει η αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως θα αντιδρασει η μηχανια αλλα αυτο δεν σημαινει πως θα πρεπει να πάμε σε ε, τόσο χαμηλές τιμές. Νομίζω πως ε, καλός είναι ο συμβασμός που έχουμε επιτύχει και νομίζω κυρία Λιχτεμπέργκερ έχουμε επιδείξει πως είμαστε σε θέση να συμβιβαστούμε σε ένα επίπεδο το οποίο είναι ρεαλιστικά εφαρμόσιμο. Αυτό είναι σημαντικό. Εγώ προέρχομαι από χώρα στην οποία βεβαίως ξέρετε δεν υπάρχουν τέτοια όρια, οπότε δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω με ε, αυτό το όριο ταχύτητας, ε, αλλά νομίζω πως γενικά είναι σημαντικό για το περιβάλλον αυτό το οποίο είχαμε στο παρελθόν με αυτό το οποίο είχε πει η Αν να χρησιμοποιηθούν έξυπνα συστήματα που μπορούν να συνεισφέρουν στην προστασία του περιβάλλοντος με το να αποφεύγουμε τα μποτιλιαρίσματα και να υπάρχει μια καθοδήγηση των ροών μέσω ορίων ταχύτητας. Αυτό νομίζω είναι σημαντικό. Αλλά γενικά καλό είναι νομίζω να θέσουμε και εμείς προδιαγραφές ως Επιτροπή Κύριε να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Βλάσακ για το ότι έχουμε εδώ πέρα μια ρεαλιστική και εφαρμόσιμη οδηγία τουλάχιστον όσον αφορά το πώς το βλέπουμε εμείς ως Επιτροπή Μεταφορών. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε πως ε, τα δύο τρίτα αυτών των οχημάτων που κινούνται στην Ευρώπη ανήκουν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μιλάμε εδώ πέρα για χειρόνακτες. Και πρέπει αυτοί οι άνθρωποι εργάζονται στο τσακ. Πράγματι όσον αφορά το χρόνο και ο κύριος ε, Στέρξε καλά είπε πως η διάρκεια ζωής των κυμάτων είναι δεκαετής και αν πράγματι και εδώ πέρα εδώ έχουμε ένα μεγάλο μπλεκ που θέλουμε να εγκρίνουμε όσον αφορά την μείωση των εκπομπών, εάν θέλουμε να οδηγηθούμε σε μία νέα γενιά κινητήρων εσωτερικής ε, καύσης, χρειαζόμαστε αυτά τα 10 χρόνια για να μπορούν επίσης και να κάνουν οι επενδύσεις α, αυτή, την, ε, οι μικρές επιχειρήσεις αυτή την επένδυση και να μην τους λέμε «Α, το πράσινο το σηματάκι που έχετε σήμερα από αύριο δεν ισχύει, θα πληρώνετε 5 ευρώ να μπαίνετε στο κέντρο της πόλης και τα λοιπά και τα λοιπά. Για να φτάσουμε στα 135. Γι' αυτό νομίζω πως η χρονική αυτή ακολουθία είναι πολύ σημαντική. Ερχόμαστε σε ένα επίπεδο που είναι κατά μέσο όρο 202 γραμμάρια. Και θα πάμε μέχρι το 2014 στα 175 και λέμε πως ένα λίτρο σημαίνει 202 ε, γραμμάρια ανά 100 χιλιόμετρα και λέμε μέχρι το 2014 κατά μέσο όρο θα πέσει άλλο στα 8 λίτρα καυσίμου και στο 2022 θα έχουμε πέσει στα 6 λίτρα κατά μέσο όρο αν το δούμε αυτό συνολικά, το πώς η εξοικονόμηση θα έχουμε σε διοξείδιο του άνθρακα είναι τεράστια. Και είναι νομίζω σωστό αυτό. Το ερώτημα τώρα, το οποίο βεβαίως εδώ πέρα πρέπει να δούμε και ποια είναι η ευθύνη των μηχανικών, τι θα γίνει στο μέλλον με τους νέους κινητήρες εσωτερικής καύσης, εάν υπάρχει μεγαλύτερη πίεση Δηλαδή όσον αφορά τα σωματίδια, το πώς θα πάμε σε μια γενιά Euro 6 όσον αφορά τις εκπομπές. Μήπως θα έχουμε μια αντίστροφη τάση και εξέλιξη, δηλαδή εάν έχουμε τα φίλτρα τα οποία δεν θα είναι όπως είναι τώρα, αλλά θα έχουμε μια πλήρη καύση. όσον αφορά τους εσωτερικούς κινητήρε, χρειαζόμαστε άρα περισσότερο καύσιμο φοβάμαι και περισσότερο ιδιοξείο του άνθρακα. Μήπως λοιπόν το Euro 6 δυσκολεύσει την εφαρμογή του Euro 5. Αυτό είναι και το ερώτημά μου προς την Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Τικάου. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ξεκινήσω λέγοντάς σας ότι στα τέλη του 2007 η δέσμη μέτρων για την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια εγκρίθηκε και βασικός στόχος της δέσμης αυτής ήταν να θέσει ξεκάθαρους στόχους για τη μείωση των εκπομπών τόσο για τον βιομηχανικό τομέα και εδώ πέρα μιλάμε για το σύστημα ανταλλαγών αδειών εκπομπής αλλά και για άλλους τομείς ιδίως για τις κατοικίες και για τις μεταφορές. Το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη έχει δεσμευτεί με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και με προθεσμία το 2020 σημαίνει ήδη ότι έχουμε μπροστά μας μια πραγματικότητα, ένα πραγματικό σημείο κίνησης. Τώρα, όσον αφορά τις συμβαστικές τροπολογίες. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να αναλύσουμε προσεκτικά το κείμενο, την έκθεση αυτή λοιπόν, από τη σκοπιά της προσφοράς, δηλαδή πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα οχήματα, τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, χωρίς να ξεχνάμε όμως και την άλλη πτυχή, την σκοπιά της ζήτησης. Γι' αυτό το λόγο υπέβαλα τροπολογίες με τις οποίες ζητώ να υπάρχουν τα απαραίτητα χρηματοοικονομικά κίνητρα προκειμένου να ενθαρρύνουμε την αντικατάσταση των παλαιών οχημάτων που ρηπαίνουν περισσότερο με νέα οχήματα, πρόσφατα οχήματα τα οποία ανταποκρίνονται στους στόχους του κειμένου. Όσον αφορά την προσφορά, εδώ πέρα μπορούμε να μιλήσουμε για την προσαρμογή των οχημάτων. Θα πρέπει να βελτιωθούν τα ελαφρά οχήματα από τεχνολογικής πλευράς προκειμένου να ρηπαίνουν λιγότερο, προκειμένου να εκπέμπουν λιγότερο διοξίδιο του άνθρακα. Οι κατασκευαστές μας λένε ότι χρειάζονται 7 χρόνια από τη στιγμή που θα αρχίσει η σύνταξη, αν θέλετε, ε, Μάλλον χρειάζονται 7 χρόνια για να κατασκευαστούν τα οχήματα αυτά, για να επινοηθεί το νεαυτό όχημα, να σχεδιαστεί και να γίνει πραγματικότητα. και χρειάζονται επιπλέον πέντε χρόνια για να παράγουν το όχημα και για να προωθηθεί αυτό στη συνέχεια στην αγορά. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε εμείς και τα απαραίτητα χρονικά στάδια για να επιτύχουμε στην πράξη αυτούς τους στόχους. Γιατί μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να κάνουμε πραγματικότητα τους φιλόδοξους αυτούς στόχους. Προσωπικά δεν νομίζω ότι τα όσα προβλέπονται αυτή τη στιγμή αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κίνητρο για τους κατασκευαστές και νομίζω ότι θα ήταν καλό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γενικότερα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δείξουν μια κάποια συνέπεια, μια κάποια συνοχή. Μια συνέπεια σε σχέση με την υφιστάμενη νομοθεσία στον τομέα των οχημάτων. Ελπίζω ότι η έκβαση όλης αυτής της διαδικασίας θα είναι θετική και ότι θα μας επιτρέψει να μειώσουμε τελικά τους ρήπους, τις εκπομπές διοξείου του άνθρακα το συντομότερο δυνατό, θα πρέπει όμως σε κάθε περίπτωση να θέσουμε στόχους ρεαλιστικούς και το χρονοδιάγραμμά μας να είναι ρεαλιστικό. Ολοκληρώνοντα, θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε χρηματοοικονομικά κίνητρα προκειμένου να αυξηθεί και η ζήτηση γιατί μπορούμε να έχουμε ένα πολύ καλό νομοθετικό κείμενο με πάρα πολύ καλούς και φιλόδοξους στόχους, αλλά δεν καταφέρουμε να ενισχύσουμε την ζήτηση για αυτά τα πιο οικολογικά οχήματα, η οδηγία δεν θα καταφέρει να πετύχει τους στόχους της. Θα ήθελα να συγχαρώ τον συντάκτη της γνωμοδότησης, καθώς επίσης και τους κοιόδης ε, εισηγητές, για όλες τις προσπάθειες που κατέβαλαν. Σίγουρα το ζήτημα δεν είναι εύκολο, αλλά είμαι σίγουρος ότι το αποτέλεσμα θα είναι πολύ θετικό. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι εύκολα τα πράγματα, γιατί υπάρχουν δύο σημαντικές πτυχές που δεν εκτιμούνται τόσο εύκολα. Πρώτα απ' όλα η τεχνολογία, γιατί έχουμε πληροφορίες τελείως διαφορετικές και εγώ θεωρώ πως αυτή τη στιγμή οι σκιώδεις ηγητές βρήκανε καλούς συμβιβασμούς, αλλά αν δούμε το τι γίνεται με την τεχνολογία μας έχει δείξει στο παρελθόν πώς πρέπει να πούμε τα, να θέσουμε ξεκάθαρους ε, στόχους και αν θέλουμε να επιτευχθεί ένας στόχος ε, αν ε, είναι κάτι το εθελοντικό δεν επιτυγχάνεται. Αν λέμε πρέπει να επιτευχθεί τότε ε, επειδή χάνεται και αυτό γίνεται για μια φορά γρηγορότερα από τις αποφάσεις που λαμβάνονται εδώ πέρα μέσα στο Κοινοβούλιο. Δεύτερον, που είναι η πολιτική μας βούληση. Πρέπει να πούμε ξεκάθαρα πως μιλάμε εδώ πέρα πάρα πολύ για τα φορτηγά και για τα ελαφρά φορτηγά. Τα, αλλά ξέρετε πως η μάζα στους δρόμους είναι τα χ. Και βεβαίως εκεί πέρα είναι η ψηφοφόροι μας, γι' αυτό γίνεται πιο δύσκολη συζήτηση, γιατί αν δούμε την ποσότητα πρέπει να ασχοληθούμε με τα γιώταχη, γιατί ξεκάθαρα μαθηματικά εκεί πέρα, αυτά είναι τα περισσότερα. Το ερώτημα, υπάρχει πολιτική βούληση να το κάνουμε αυτό. Το ίδιο και για ταχύτητα. Λυπούμε. Όλοι ξέρουν πως αν πάνε πιο σιγά μειώνονται τα ατυχήματα και η κατανάλωση. Και όλες οι χώρες έχουν όρια ταχύτητας πλην ε, μίας δύο. Και πρέπει τώρα τεχνικά να δούμε το πολιτικό πρόβλημα αυτών των χωρών με το να ε, εισαγάγουμε εδώ πέρα εμείς ώρα γιατί σε κάποιες χώρες δεν έχουν το θάρρος να βάλουν όρια ταχύτητας. Ε, δεν είναι σωστό αυτό. Το καλύτερο είναι να τους πούμε, κοιτάξτε εσείς αυτές οι χώρες κάντε τη δουλειά που πρέπει να κάνετε, θα μειωθούν και τα ατυχήματα, μήπως να μειώσετε ταχύτητα. Τέλος, όσον αφορά τα, τα γεωταχή, και εγώ τα διαβάζω αυτά τα, τα φυλάδια. Αλλά γιατί να έχουμε ένα μάξι με 400 και 500 ύπους. Γιατί φτιάχνουμε ένα μάξι που πηγαίνει τόσο γρήγορα και τόσο δύσκολα ελέγχεται και είναι άσχημο και για το περιβάλλον και για την υγεία. Μήπω θα πρέπει να αλλάξει η διαφήμιση. Και ναι, εμεί να στείλουμε ένα πολιτικό μήνυμα, να πάμε σε μια άλλη κατεύθυνση, να πούμε ότι το cool αυτοκίνητο θα πηγαίνει πιο σιγά. Μεταξύ δηλαδή τεχνολογίας και πολιτικής βούλησης υπάρχει μια ψαλίδα και το δύσκολο πρόβλημα βεβαίω είναι αυτό πρέπει να λυθεί στις χώρες. Και τελευταία παρατήρηση, θεωρώ πως ε, σύν το χρόνο θα αποδειχθεί πως τα καθαρότερα οχήματα είναι και οικονομικότερα για τις εμιχειρήσεις και θα ωφεληθεί και η παραγωγή και η έρευνα στην Ευρώπη. Αλλιώς θα φτιαχτούν και θα τα εισάγουμε από την Κίνα ή από κάπου αλλού. Οπότε ας κοιτάξουμε λίγο το μέλλον, αλλά να έχουμε και λίγο περισσότερη βούληση και θάρρος για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα εκεί που πραγματικά είναι. Τρεις ακόμα μελητές. Ναι, δώσω τον λόγο στην Κομισιόν. Uh, next is Mr. Ο κύριος Bradbourne. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε να άρχισα να ακούω πολωνικά για μια στιγμή από την αγγλική διερμηνία, δεν άκουσα πολύ καλά τα πάντα. Παρακλούσα τέλο πάντων τη συζήτηση, δεν ήθελα αρχικά να πάρω το λόγο, αλλά τα όσα άκουσα, ω συνήθω ε, στην Επιτροπή αυτή, δεν έχουν μεγάλη επαφή με την πραγματικότητα. Η κυρία Τικάου έθιξε πολύ καλά το ζήτημα, να δούμε τι μπορούμε να πετύχουμε, πότε μπορούμε να το πετύχουμε και να δούμε επίσης πώς μπορούμε να αυξήσουμε και τη ζήτηση. Μόνο έτσι θα καταφέρουμε να επιλύσουμε το ζήτημα που έχουμε μπροστά μας. Συμφωνώ με τις τροπολογίες του κυρίου Βλασάκ ως προς αυτό και κατά την άποψή μου διατρέχουμε τον κίνδυνο να απομακρυνθούμε πάρα πολύ από την πραγματικότητα. Όπως είπε η κυρία Τικάου, χρειάζονται 7 χρόνια για να σχεδιαστεί μία νέα μηχανή, ένα νέο κινητήρα. μέχρι να σχεδιαστεί και να παραχθεί. Και θα πρέπει αυτό να το έχουμε κατά Δεν μπορούμε να κάνουμε εμεί τίποτα άλλο για να τα αλλάξουμε. Έτσι λειτουργούν τα πράγματα. Επομένω, γίνετε, σα παρακαλώ, πολύ ρεαλιστέ σε σχέση με του στόχου που θέτετε. Αυτό που με κάνει να θέλω να πάρω το λόγο είναι ότι γίνονται κάποιε αναφορέ, όπω για παράδειγμα το να χρησιμοποιούμε συσκευέ μείωση ή ελέγχου τη ταχύτητα. Νομίζω ότι αυτό ισχύει σε κάποιες περιοχές αλλά δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να αρχίσει να ισχύει κάτι τέτοιο στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, γιατί τα οχήματα αυτά μπορούν ή θα πρέπει τουλάχιστον να μπορούν να επιταχύνουν περισσότερο σε αυτοκινητοδρόμους. Το να μην τους δώσουμε τη δυνατότητα να επιταχύνουν και να καταφέρουν να ξεπερνάνε άλλα οχήματα όταν κυκλοφορούν σε αυτοκινητόδρομους, νομίζω θα δημιουργήσει περισσότερα ατυχήματα από ό,τι θα περιορίσει. Επίσης είπανε κάποιοι ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και ITS, ευφύ e, συστήματα μεταφορών. Δεν ξέρω αν έχετε πάει κύριε Πρόεδρε στους αυτοκινητοδρόμους γύρω από το Μπέρμιχαμ, αλλά υποτίθεται ότι έχουμε συστήματα για ευφύς μεταφορές στους δρόμους αυτούς και χθε ενώ πήγαινα στο αεροδρόμιο στις 10.30 το πρωί, άρχισε να ισχύει ένα τέτοιο σύστημα το οποίο τελικά έκανε τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα, δημιούργησε μεγαλύτερη συμφόρενση και νομίζω πραγματικά ότι δεν ωφελούν τόσο πολύ, δεν μπορούν να επιφέρουν θετικά αποτελέσματα. Επομένως, ας γίνουμε πιο ρεαλιστές, ας συνειδητοποιήσουμε τι μπορεί να παράγει η αυτοκινητοβιομηχανία και ας ξεκινήσουμε να νομοθετούμε με αυτή τη βάση. Ήμουνα στο αυτοκινητόδρομο M6M5 το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και όντως και εγώ έκανα πάρα πολύ ωραία, έμπλεξε και πέρασε συμφόρηση. Ναι, να περάσετε από τα διόδια όμω τότε, λέει ο κύριο Μπράντμπουρν. Ναι, αλλά αυτό δεν με βόλευε για να πάω στο Κάρντιφ. Ο κύριο Χίγκινγκ έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτά που είπε ο κύριο Κούν, Πικέ και Μπράντμπουρν και να ευχαριστήσω και τον ε, εισηγητή, ο οποίος πιστεύω ότι έχει απόλυτο δίκιο. Θα πρέπει να πετύχουμε την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στην περιβαλλοντική πτυχή και την εμπορική πτυχή θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι αυτοκινητοβιομηχανίε είναι ένα πολύ σημαντικό εργοδότη στην Ευρώπη και χάνουμε ήδη πάρα πολύ μεγάλο μερίδιο τη αγορά σε σχέση με την Κίνα, για παράδειγμα. Επίση, στα πλαίσια τη ε, οικονομική κρίση υπάρχουν πολλοί εργοδότε οι οποίοι θα χάσουν μερίδιο τη αγορά και θα μπορούν να προσλαμβάνουν αν αρχίσουμε να επιβάλλουμε τους περιορισμούς που προβλέπονται. Επομένως, πιστεύω ότι οι συμβαστικές τροπολογίες πετυχαίνουν πάρα πολύ καλά την ευκταία ισορροπία. Επίσης, όσον αφορά την ε, εξαίρεση από το... μέχρι τις 25.000. Αυτό ήταν πολύ θετικό. Επίσης, συμφωνώ με την πρόταση που γίνεται για τα πρόστιμα, τη μείωση των προστήμων. Και αυτό που βλέπουμε πολύ συχνά είναι όταν μειώνται τα πρόστιμα, τότε εφαρμόζονται τελικά. Και νομίζω ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να βελτιώσουμε και τεχνολογία και να παράγουν ε, τα αυτοκίνητα λιγότερε εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα. Το σημαντικό επίση να δούμε ποιο θα είναι το σύστημα εποπτεία. Γιατί α, τα πράγματα θεωρητικά είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά όταν πρέπει να εφαρμόσουμε ένα σύστημα εποπτεία στην πράξη, τα πράγματα κάπω δυσκολεύουν. Επίση, να συμφωνήσω και με την κυρία Τικάο στην πρόταση που έκανε για να βγάλουμε εκτός κυκλοφορίας τα παλαιά οχήματα. Ένα από τα λογικά πράγματα που έχουμε κάνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν το να δημιουργήσουμε ένα σύστημα το οποίο προβλέπει οικονομικά κίνητρα προκειμένου να αποσύρονται τα παλαιά οχήματα και να μπορούν οι ε, οδηγοί να τα αντικαθιστούν πιο εύκολα με νέα οχήματα. Νομίζω λοιπόν ότι ε, είναι πολύ σημαντικές προτάσεις που γίνονται εδώ πέρα θα ήθελα να συγχαρώ τον συντάκτη της νομοδότησης για τις πολύ καλές συμβαστικές τροπολογίες οι οποίες κατέληξε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν ήθελα στην αρχή να παρέμβω. Όλοι μας λάβαμε πληροφορίες ε, για διάφορα βιομηχανικά για να δούμε που ήταν τα όρια και οι ημερομηνίε, οι προθεσμίες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πρόβλημα. Εδώ Θέλεις όμως να παρέμβω για τα μηχανήματα που περιορίζουν την ταχύτητα. Εδώ στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή βλέπουμε ότι δημιουργείται μια συζήτηση πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα και με τα κράτη-μέλη που είναι ιστορικά κατά του περιορισμού της ταχύτητας και σε όλους τους δρόμους και έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν έτσι. Να αυτή τη φορά για την ε, ασφάλεια την οδική, αυτό είναι το ηρωνικό τώρα, και για το περιβάλλον, για την προστασία του. Να που μπορούμε να θέσουμε το θέμα έτσι και με διάφορες ορισμένες χώρες για τις οποίες και μιλάμε που έχουν ε, την τεχνολογία και ε, κατά ανταγωνιστικό τρόπο και το να είναι κανείς υπέρ αυτών ε, των μηχανημάτων που περιορίζουν ταχύτητα σαν μια καινοτομία τεχνολογική που βοηθάει και την προστασία του περιβάλλοντος ε, και την ασφάλεια είναι κάτι θετικό. Όπως και ο συνάδελφος ε, δεν ξέρω αν θα έπρεπε να τρέξουμε τόσο αλλά θα πρέπει να το θέσουμε αυτό σαν θέμα. Γιατί δρόμους μιλάμε και εκεί που υπάρχουν ουρές αριστερά-δεξιά ακριβώς οχημάτων και ποιοι θα πρέπει να είναι γρήγοροι δρόμοι κλπ. Θα μπορούσαμε έτσι να απλοποιήσουμε και είμαι υπέρ της τοποθέτησης του θέματος κατά τον τρόπο αυτό. Επίσης από την Επιτροπή συμφωνώ απόλυτα ότι η συμβαστική λύση αν μπορεί να προχωρήσει εντάξει είμαι υπέρ αλλά αντιμετωπίζω εδώ το θέμα εδώ για τα την οργάνωση αυτών των αυτοκινήτων για την ασφάλεια των επιβατών. Έχουμε το συζήτηση αυτή με τη βιομηχανία, κάτι το ρεαλιστικό και κάτι από την άλλη μεριά κάτι το φιλόδοξο. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε με την Επιτροπή και λοιπά μήπως καμιά φορά ε, σιωπούμε ε, για ρεαλισμό. Δεν ξέρω αν έχουμε ε, και μια γυάλινη σφαίρα για να δούμε τα πράγματα, να τα προβλέψουμε, μήπως υπάρχουν και άλλοι και είναι περισσότερο ανταγωνιστικοί για να είμαστε εμείς ρεαλιστές με αυτή τη βιομηχανία. Τελικά τους κάνουμε χάρες και δεν τους παροτρύνουμε για να είναι περισσότερο ανταγωνιστικοί. Γι' αυτό παρακαλώ οι στην Επιτροπή να μας διαβεβαιώσουν ότι δεν χάνουμε έδαφος με τη βιομηχανία, με τις συμβαστικές αυτές λύσεις. Ευχαριστώ. Σαλονίτση από πλευράς Επιτροπής. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σε όλους. Καταρχάς να κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα όσον αφορά τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα βασίζεται σε μια μελέτη αντικτύπου και σε τεχνικές μελέτες οι οποίες κατέληξαν στο ότι η πρόταση αυτή, καθώς επίσης και η βραχυπρόθεσμη και η μακροπρόθεσμη στόχη της, είναι λογική. Επομένως, θεωρούμε ότι με τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Όσον αφορά τις ε, προτινόμενες συμβαστικές τροπολογίες που συζητήσατε σήμερα, καθώς επίσης και τα σχόλια που έγιναν για τους ε, στόχους ε, των 175 και 135 γραμμαρίων διοξιδίου του άνθρακα, και πάλι θεωρούμε ότι η δική μας πρόταση είναι η καλύτερη. Όσον αφορά την συμβαστική τροπολογία Γ, θα ήθελα να πω ότι όπως υπόθηκε ήδη, ότι τα 95 ευρώ αναγραμμάριο δεν ευθυγραμμίζονται με το κόστος το οποίο προβλέπεται για την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών. Επομένως δεν είναι αυτό ένα ιδανικό πρόστιμο το οποίο θα μας βοηθούσε να πετύχουμε τον στόχο μας. Ο περιορισμός της ταχύτητας και η συμβαστική τροπολογία Β, που είναι και η πιο ευαίσθητη από ό,τι κατάλαβα, είναι πολύ σημαντικό να δούμε αν η προτινόμενη τροπολογία μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη. Αυτή τη στιγμή δεν είναι σαφές αν αυτά τα τρία γραμμάρια διοξιδίου του άνθρακα ανά 10 χιλιόμετρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημείο αναφοράς και αν πραγματικά η εξήγηση που δίνεται είναι σωστή. Θα πρέπει να δοθεί μια εξήγηση ή δυνατόν μέσω με κάποιας μελέτης. Ευχαριστούμε. Κύριε Βλασάκ, θέλετε να προσθέσετε εσείς κάτι. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να σας πω ότι άκουσα κάποιες ε, πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις. Όλοι πλέον ξέρετε ποια επιχειρήματα, ποιες ιδέες είναι πιο σχετικές με το ζήτημα και ποιες όχι. Ας ξεκινήσω με αυτό που είπα στην αρχή της παρεμβασής μου. Πιστεύω ότι ε, η τοποθέτηση της Επιτροπής των Μεταφορών θα πρέπει να ασχολείται με τεχνικά ζητήματα, με ζητήματα που άπτονται των μεταφορών και ότι ε, θα πρέπει κατά αυτόν τον τρόπο να συμβάλλουμε εμεί προς την Επιτροπή Περιβάλλοντο, η οποία με τη σειρά τη είναι αρμόδια γιατί ό,τι έχει να κάνει με τι εκπομπέ. Και έχω μία αντίρρηση στο σημείο αυτό. Εκτιμώ ιδιαίτερα την ε, συζήτηση που έλαβε χώρα, καθώς επίσης και τις που γίνανε για την ε, διαπραγμάτευση της γνωμοδότησης αυτής, αλλά διαφωνώ με αυτό που υπόθηκε ότι η Επιτροπή μας αποτελεί ε, τροχοπέδι στις ε, εξελίξεις που θέλουμε να πετύχουμε και στην πρόοδο που θέλουμε να σημειώσουμε. Σε καμία περίπτωση σύμφωνο με αυτό. Όσον αφορά τώρα με τους μηχανισμούς, τα όργανα περιορισμού της ταχύτητας. Κοιτάξτε, έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες όσον αφορά την λειτουργία των, των μηχανισμών αυτών, την ασφάλεια, το αν μπορεί κανείς να προσπεράσει εύκολα ένα άλλο αυτοκίνητο, στο αν οδηγούν σε μείωση γενικότερα της ταχύτητας στους αυτοκινητοδρόμους, στο πώς μπορούν να εφαρμοστούν στα πλαίσια μιας εθνικής νομοθεσίας και όσον αφορά και το κόστος χρησιμοποίησής τους τα νέα οχήματα θα έχουν το μηχανισμό αυτό, αλλά αν τα παλιά οχήματα πρέπει να εξοπλιστούν με τη σειρά τους, τότε αυτό θα οδηγήσει σε μεγαλύτερο κόστος. Επίσης κάποιος θα πρέπει να εποπτεύει όλη αυτή την κατάσταση. Δεν είμαι κατά των ε, περιοριστών ταχύτητας, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε το ζήτημα αυτό σε μια ξεχωριστή έκθεση και να ισχύει το σύστημα αυτό για όλα τα οχήματα εν γέννη. Αυτό άλλωστε είχα πει και στην αρχή της παρέμβασής μου. Και το ζήτημα ουσιαστικά αυτό βρίσκεται στο περιθώριο, αν θέλετε, του βασικού ζητήματο το οποίο πρέπει εμεί να συζητήσουμε. Σα ευχαριστώ πολύ για τη σύντηση αυτό, αυτή και ελπίζω θα λάβουμε τη σωστή απόφαση αύριο. Σα ευχαριστώ κύριε Βλασάκ. Συμφωνώ μαζί σα. Η Επιτροπή μα δεν είναι αρμόδια για περιβαλλοντικά ζητήματα. Και επίση πολλέ φορέ εμένουμε πάρα πολύ σε κάποιε αρχέ, αλλά δεν προχωρούμε γρήγορα στι πράξει. Ψηφίζουμε αύριο στην Επιτροπή μας, θα γίνει το Σεπτέμβριο ψηφορία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και στην Ολομέλεια η έκθεση αυτή θα πάει τον Νοέμβριο του 2010. Σας ευχαριστώ πολύ όλους για τη συζήτηση. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή σχετικά με τους σαρωτές σώματος. Ξέρω ότι ο κύριος Ρόιτε είναι εκτός αιθούσης. επομένω θα τον προσκαλέσουμε να μπει στην αίθουσα. και ζητήσαμε και από κάποιους συνοδέλφους της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών να έρθουν εδώ Ξέρω ότι θα είστε πολλοί αυτοί οι οποίοι θέλετε να πάρετε το λόγο, αλλά μην το κάνετε αυτό τώρα. Θα σας πω ποια στιγμή, στιγμή να σηκώσετε τα χέρια προκειμένου να σας γράψω όλους τον κατάλογο των ομιλητών. Vice President as well. Okay, so those who want to speak, you can start to indicate now and the Secretary. Λοιπόν, μπορείτε πλέον να πείτε στη γραμματεία ότι θέλετε να πάρετε το λόγο. Έχουμε πάνω κάτω μία ώρα, επομένως αν 65 ομιλητέ, δεν χρειάζεται να είναι κανείς ε, genius στα μαθηματικά για να καταλάβει πόσο χρόνο τον αλογεί. Κύριε Ρόιτε, έχετε το λόγο. Thank you very much, Chairman. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είναι ευχαρίστηση να επιστρέφω στην Επιτροπή σας μετά την τελευταία φορά που συζητήσαμε τις προδιαγραφές ασφαλείας τον Ιανουάριο. Τέλος Ιανουαρίου υποσχέθηκα εξ ονόματος Κομισιόν μια έκθεση από το Μάρτιο-Απρίλιο και ζητώ συγγνώμη γιατί έχει πάει 15 Ιουνίου αλλά νομίζω θα συμφωνήσετε πως η τέφρα η φεστιακή δυσκόλεψε τα πράγματα. Οπότε να σας πω έτσι λίγο γρήγορα τα της έκθεσης ε, εξ ονόματος του Αντιπρόεδρου της Κομισιόν του κυρίου Κάλας Ήταν πολύ καλή, καλός συντονισμός γιατί ήθελε ε, να δείτε την έκθεση πριν την συζητήση με τους Υπουργούς Μεταφορών την Πέμπτη. Λοιπόν, τώρα το πλαίσιο της έκθεσης είναι σαφές σχετικά. Έχουμε έναν κανονισμό ασφαλείας, τον οποίο επεξεργαστήκαμε από κοινού, είναι ο 208. Και θα θυμάστε πως είχαμε εφαρμοστικά μέτρα το 2008. Το δεύτερο μέρος, το το δεύτερο μισό του έτους. Μας ε, δείξατε τότε την κίτρινη κάρτα όσον αφορά όλα τα μέσα που έχετε στην διάθεσή σας ε, για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια στα αεροδρόμια. Δεν είμαστε σίγουροι για ένα πράγμα τότε, αυτό το οποίο λέγαμε σαρωτές σώματος, οπότε τελικά το αφαιρέσαμε και υποσχεθήκαμε να επανέλθουμε με μια έκθεση. Αυτή είναι λοιπόν η έκθεση που έχετε μπροστά σας έκθεση η οποία πρέπει να λάβει υπόψη και κάποιες ατυχείς ε, συνθήκες, ε, τώρα δεν θα αναφέρω. Ξέρετε, την πτήση της Northwest ε, και την επιπλέον απειλή ε, τρομοκρατίας στις αεροπορικές μεταφορές. Ποια είναι η κατάσταση. Τα γεγονότα. Τα γεγονότα είναι πως έχουμε κράτη-μέλη που χρησιμοποιούν σαρωτές σώματος, Φιλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία, Γαλλία, Ιταλία. Η Ιταλία το σκέφτεται. Έχουν μια κατάσταση ανά τον κόσμο όπου χρησιμοποιούνται αυτοί οι σαρωτές, Είπα Καναδάς, δεν θα τα αναφέρω αυτά, αυτά αναφέρονται στην έκθεση. Οπότε το πρώτο ερώτημα είναι, είναι νόμιμο κάτι τέτοιο. Η απάντηση είναι ναι, σύμφωνα με τους υπάρχοντες κανονισμούς, γιατί μπορούμε να έχουμε περαιτέρω μέσα έρευνας, ε, είτε πιο αυστηρά, είτε αν θέλει κανείς να κάνει κάποιο πείραμα. Και από αυτές τις διατάξεις λοιπόν τις δύο του κανονισμού μπορεί να γίνει χρήση των σαρωτών και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα είναι, θέλουμε να γίνει αυτό όπως γίνεται αυτή τη στιγμή, με το κάθε κράτος μέλος να έχει τους δικούς του κανόνες ή καθόλου κανόνες όσον αφορά την χρήση αυτών των πραγμάτων και θέλουμε να αμφισβητήσουμε την ασφάλεια σε μία μόνο ε, στάση. Νομίζω λοιπόν πως η έκθεση τα λέει λεπτομερώς και ικανοποιητικά. Κάποιες απαντήσεις τώρα στις πρώτες ερωτήσεις, τις ερωτήσεις κλειδιά που κάνατε. Πρώτα απ' όλα ερώτηση κλειδιά της, κλειδί της αποτελεσματικότητας. Δεύτερο ερώτημα υγεία. Τρίτο σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και τέταρτον κόστος και όφελος. Ε, θα είμαι σύντομος γιατί δεν νομίζω πως έχει νόημα να μπω στις λεπτομέρειες. Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, η έκθεση καταδεικνύει πως πολλά κράτη-μέλη και η Κομισιόν θεωρούν πως ε, οι νέου τύπου σαρωτές μπορούν να είναι ένα αποτελεσματικό μέσο ανείχνευσης εκρηκτικών που δεν είναι μεταλλικά ε, και που είναι κολλημένα στο σώμα. Ε, δεν υπάρχει εγγύηση 100%. Είναι σαφές αυτό, μπορούμε να το πούμε. Αλλά θα είναι πιο αποτελεσματικός άνεχος εξετάζουμε τις τέσσερις διαφορετικές τεχνολογίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά όσον αφορά τους αρωτές ασφαλείας παθητικών και ενεργητικών μικροκυμάτων ε, ακτίνων ε, ρέντγεν και των δύο τεχνολογιών. Ε, δεν έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή βγάλουμε κάποιο αποτέλεσμα, αλλά από ό,τι φαίνεται οι εθνογραφίε δεν χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξετάζουμε λοιπόν το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι το μεγάλο θέμα. Ήταν το μεγάλο θέμα πριν από 1,5 χρόνο. Και καταλήξαμε πως υπάρχουν τεχνολογίες τις οποίες τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν είναι τόσο ακανθώδη, θα έλεγα πως μπορούν να αντιμετωπιστούν κιόλα. Δηλαδή στον πάρο προστασία δεδομένων, αξιοπρέπεια, εισβολή στην ιδιωτική σφαίρα, προστασία της οικογένειας, υπάρχουν πολλά ζητήματα που έχουν αναφερθεί. Το θέμα είναι υπό ποιους όρους χρησιμοποιείται αυτή η τεχνολογία και πώς θα διασφαλίσουμε πώς ε, είναι, αν θέλετε, ουδέτερη ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα αυτή η τεχνολογία. Τρίτον, το τέταρτο μάλλον, ε, είναι το θέμα κόστους και ωφέλους που αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι το δύσκολο, μια δύσκολη ανάλυση μπορούμε να πούμε πως υπάρχουν κάποια στοιχεία για μείωση του κόστους και όλες. Οπότε, συμπερασματικά για εμάς το ζήτημα είναι τι κάνουμε τώρα. Αλλά τα όλα να είμαι σαφής. Αυτή η στιγμή η κατάσταση είναι ως εξής. Η τεχνολογία αυτή αναπτύσσεται στην Ε, χρησιμοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς κοινούς κανόνες με διαφορετικές ε, προσεγγίσεις. Οπότε το ερώτημα είναι μήπως θα έπρεπε να ορίσουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης κανόνες που αφορούν την προστασία της υγείας των επιβατών αλλά και του προσωπικού των αεροδρομίων. Μήπως θα έπρεπε να ορίσουμε τους κανόνες για την διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. και βεβαίω αυτό θα γίνει στο πλαίσιο του κανονισμού 300-208 γιατί έχουμε όλα τα άλλα μέσα να κάνουμε γιατί όλα τα άλλα μέσα ούτως ή άλλως ρυθμίζονται δηλαδή οι σκύλοι, οι ανιχνευτές μετάλλων, όλα αυτά αλλά ακόμα και αν κάναμε κάτι τέτοιο να είμαι σαφής θα είναι μόνο μία επιλογή μεταξύ άλλων για τα κράτη-μέλη. Οπότε αν έχουμε ένα σαρωτή ως ένα μέσο ανείχνευσης στην οδηγία την εφαρμοστική του κανονισμού, δεν θα λέει πως τα κράτη-μέλη πρέπει να χρησιμοποιήσουν σαρωτή. Μετά, όταν ένα κράτος μέλος ε, το έχει χρησιμοποιήσει, να δούμε την ε, επιλογή του πράγματος. Αλλά εάν δούμε το σκεπτικό της έκθεσης προς τα εκεί πάει σαφώς, γιατί γνωρίζουμε την πολιτική ευαισθησία, οπότε η Κομισιόν θα ακούσει το Κοινοβούλιο, θα ακούσει τα κρατημέλη όσον αφορά τη συζήτηση αυτής της έκθεσης και μετά με βάση αυτή τη συζήτηση θα έχουμε κάποια μορφή εφαρμοστικής νομοθεσίας αν πάει προς αυτή την κατεύθυνση αλλά σαφώς όχι χωρίς να έχει γίνει μια λεπτομερής αξιολόγηση αντικτύπου. Προσπάθησα να είμαι σύντομος λοιπόν, ε, κύριε Πρόεδρε, για να δεχτώ και ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε κύριε Ρόιδε που ήσταν σύντομος. Κατά αυτόν τον τρόπο δίνουμε τη δυνατότητα και στους συναδέλφους που είναι πολλοί να θέσουν ερωτήσεις. Δεκαπέντε είναι ομιλητές αυτή τη στιγμή. Θα κλείσω κατάλογος και θα πρέπει να ακολουθήσετε ένα, μια πειθαρχία. Γκρός, Αλκαντράουι, Μάισνερ, Λίχτενμπέργκερ, Φώστερ. Λάτφορντ, Βαν Όρντεν, Δε Γκράντες Πασκουάλ, Λάιτφριντ, Βαντάλεν, αυτοί είναι ομιλητέ λοιπόν. Προτείνω να κλείσω ο κατάλογο ομιλητών. Υπάρχει κάποιο που θέλει να μιλήσει, αν ναι, πείτε το τώρα, διαφορετικά δεν θα σα δώσω τη δυνατότητα αργότερα. Κυρία Τικάου, μάλιστα. Σαν δημοπρασία είμαστε εδώ πέρα. So that's it. Going, going Άλλος κανείς. Κύριε Ρικέ, σας έχουμε συμπεριλάβει, ναι. Okay, right, Έκλεισε ο κατάλογος. Πολύ ωραία. Δεν υπάρχει λόγος να σηκώσετε πλέον το χέρι σας. Δεν θα μπείτε στον κατάλογο. Έχετε δύο λεπτά ο καθένας και ξεκινάμε με τον κύριο Γκρός. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και τον πρόσωπο της Κομισιόν. Σύντομα, Σημαντικό είναι να πούμε πως πρέπει να βελτιωθεί η ασφάλεια, αλλά 100% ασφάλεια δεν υπάρχει, οπότε το ερώτημα είναι εάν θα πρέπει να εισαχθεί αυτό παντού στην Ευρώπη. Όχι, αλλά εάν εισαχθεί τότε θα πρέπει να υπάρχουν κάποια κριτήρια. Και το ερώτημά μου είναι, η Κομισιόν είναι σε θέση να δώσει τεχνικές οδηγίες, π.χ. για αμοιβαία αναγνώριση μεταξύ των χωρών και ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την υγεία, δεύτερον όσον αφορά διαχείριση δεδομένων, ιδιωτική ζωή κτλ. Γιατί νομίζω πως αναμένουμε κάποιες οδηγίες από την Κομισιόν και ξεχνάμε βεβαίως τα υγρά, το οποίο επίσης δεν έχει λυθεί γιατί πάμε από τη μία έρευνα στην άλλη και κανένα πρόβλημα δεν λύνεται. Οπότε είναι συνολικό το πακέτο. Τέλος, ε, σε διεθνές επίπεδο ποια είναι η λύση. Μήπως ε, θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε σε μια κατάσταση στην οποία ένα αεροδρόμιο θα αντιδρά με τρόπο ώστε να κάνει καψόνια στους ε, επιβάτες. Αυτά από μένα κύριε Πρόεδρε και ελπίζω να είμαι σύντομος. Πράγματι, ένα λεπτό και 45 εξαιρετικά. Κύριε Αλχαντραούι και εσείς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον εκπρόσωπο της Νομίζω πως ε, το συνολικό συμπέρασμα που βγαίνει από το έγγραφα είναι πως χρειάζεται μία εναρμονισμένη ευρωπαϊκή ε, προσέγγιση και εδώ πέρα συμφωνώ. Κάποια κράτη-μέλη δεν περίμεναν, ανέλαβαν πρωτοβουλίες. Φαίνεται πως βεβαίως αυτό ήρθε σε μία... Ε, έστω και αν είναι ε, υποπροσωρινή μορφή με τα τεστ ε, τα οποία προβλέπονται, τα οποία από την νομοθεσία περιορίζονται σε 30 μήνες ή ως συμπληρωματικά μέσα, αλλά τότε χωρίς να αντικαθιστούν τις υπάρξεις διαδικασίες, αλλά επιπλέον. Οπότε το ερώτημα είναι τι θα γίνει όταν περάσουν αυτοί οι 30 μήνες. Θα ξεκινήσουν κάποιες διαδικασίες για να ρυθμίσει με αυτό το πράγμα νομοθετικά ή να το σταματήσουμε, πώς θα γίνει. Δεύτερον, φαίνεται ότι δεν ξεφορτωνόμαστε αυτό που λέει ο κύριος Λάχτη για τη χρηματοδότηση αυτών των μέτρων ασφαλείας, γιατί ξέρετε πως κλασικά τα κράτη-μέλη τα οποία πηγαίνουν παραπέρα από ό,τι ορίζουν οι κανονισμοί πληρώνουν από μόνο τους. Και τέλος, Δεν θέλω εγώ να πω τι μορφή θα πρέπει να έχει ένας τέτοιο ευρωπαϊκός κανονισμός, αλλά συμφωνώ με αυτό το οποίο λέτε. Δεν επιτρέπεται να πούμε πως όλα τα αεροδρόμια θα πρέπει να έχουν αυτό το σύστημα, αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε τεχνικές προδιαγραφές έτσι ώστε να, έχει τη δυνατότητα, να έχουν δυνατότητα οι άνθρωποι να περάσουν ή να αρνηθούν να περάσουν από ένα σαρωτή και να υπάρχουν κάποιες εναλλακτικέ. Ε, αυτά νομίζω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Αλχαντραγουή. Ένα 58. Η κυρία Μάισνερ κατόπιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν πολλά επιχείρηματα υπέρ. Με αυτά θα ξεκινήσω. Υπάρχουν κάποιοι που, μάνατζερ που λένε εγώ δεν θέλω να περιμένω. Δεν ε, έχω κανένα πρόβλημα να περάσω. Αυτό είναι υπέρ. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τόσες ασφάλειες θα μπορούσαμε να έχουμε. Και θα είχαμε επιτύχει αυτή την ασφάλεια αν ελέγχαμε και τα υγρά και τις αποσκευές. Υπάρχουν κάποια κρατημέλη που τα χρησιμοποιούν και δεν έχει νόημα, όπως λέει και ο κ. Καντράου, να κάνω ο καθένας ό,τι θέλει. Δεν μιλάμε για ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό, έτσι. Κατά τώρα, υπάρχουν πολύ περισσότερα επιχειρήματα. Ποτέ θα έχουμε 100% ασφάλεια. Μπορούμε να δούμε μόνο το εξωτερικό και όχι το εσωτερικό του σώματος. Αυτό γίνεται μόνο με ακτίνες ρέντγεν. Υπάρχουν ιατρικές αμφιβολίες επίσης. Προστασία δεδομένων. Ποιος βλέπει τι, τι παράγεται ως εικόνα και πού αποθηκεύεται. Ε, κάτι το οποίο είδαμε στην αντιπροσωπεία στη ΣΥΠΑ δεν θέλουμε να το δούμε στην Ευρώπη, αν έχουμε δηλαδή μόνο ένα πράσινο OK. Υψηλό κόστος. Ποιος πληρώνει. Είπατε πως πρέπει να το κάνουν τα κράτη-μέλη επίσης βάρος με τα σαρωτές ε, αποσκευών. Μετά καταναγκαστικά ε, μέτρα, δηλαδή όταν αρνούνται κάποιοι μουσουλμάνοι στην ε, Μεγάλη Βρετανία αναγκάζονται να υποστούν κάτι άλλο. Και τέλος, είναι δυνατόν εάν ε, ψηφίσουμε κάτι τέτοιο να υπάρξει ένα τέτοιο κίνδυνο στην Ευρώπη, κάτι το οποίο θέλουμε. Ευχαριστώ. Η κυρία Λίχτενμπεργκερ, ευχαριστώ για την εισαγωγή στην ε, έκθεσή σας. Ε, θα ήθελα να αναφέρω κάποια ερωτήματα. Το ένα αφορά την υγεία και αν βλάπτει δεν υπάρχουν οριστικές μελέτες πώς θα μπορέσουμε να μην χρησιμοποιήσουμε ακτίνες ε, για ακτινογραφία σε ακτίνες ρέντγεν. Δεν ε, νομίζω να είναι σαφές. Ε, επίσης εγώ είμαι κάπως προσεκτική όσον αφορά την ανάλυση κόστους κόστους-οφέλους, γιατί θα πρέπει να γίνουν μετασκευές σε πολλά αεροδρόμια και αυτό κοστίζει και πρέπει να συνυπολογιστεί. Δεύτερον, το προσωπικό το οποίο δεν ξέρουμε τι, ε, εάν υπάρχει εξοικονόμηση, γιατί οι περιπτώσει αμφίβολες ούτως ή άλλως θα πρέπει να ελεγχθούν με τα χέρια και τρίτον, όπως είπε και ο κύριος Γκρό, θα πρέπει ούτως ή άλλως να το δούμε ως συνολικό πακέτο και με τους σαρωτέ υγρών, γιατί και εκεί πέρα χρειάζονται μετασκευέ στα αεροδρόμια. Και βεβαίω θα καθυστερήσουν έτσι ούτως ή άλλως οι επιβάτες και οι δύο τεχνολογίες. Ε, πρέπει να εξεταστούν. Για εμένα λοιπόν προκύπτει το εξής. Εγώ θέλω κανόνες που περιορίζουν τα πράγματα όσον αφορά την αξιοπρέπεια, την υγεία για όσους θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτή την τεχνολογία, αλλά δεν συμφωνώ με αυτόματο ε, εξαναγκασμό χρήσης αυτής της τεχνολογίας. Γιατί ε, δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, αν υπάρχει κάποιο όφελος, αν υπάρχει κάποια βελτίωση και από την έκθεσή σας δεν προκύπτει. Ε, δεν απαντάτε σε αυτά τα οποία λέμε για προστασία δεδομένων κτλ. Ε, για μένα εξακολουθούν να παραμένουν πολλά ερωτήματα ανοιχτά. Ευχαριστώ. Κυρία Φώστερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χάρη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχουμε μια καλή προσέγγιση, μόνο ότι υπάρχουν κάποια ερωτηματικά ακόμα. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι όλοι θα ήμασταν υπέρ μιας καλής προσέγγισης ασφάλειας και ελέγχου. Έχουμε βέβαια και κάποιες ανησυχίες και υπάρχουν πάρα πολλοί επιβάτες που έχουν ανησυχίες. Τώρα, ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται τώρα και που θα χρησιμοποιείται και στο μέλλον είναι ο millimeter wave. Επομένως, ε, δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Πάντως, το Ηνωμένο Βασίλειο μας ε, επιβλήθηκε ένας εξοπλισμός οπισθοσκέδασης και έχουμε κάποια παραδείγματα στον Ηνωμένο Βασίλειο με ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει συγκεκριμένε επεμβάσεις. Βλέπουμε ότι υπάρχουν μεταλλικά αντικείμενα τα οποία έχουν προσθεθεί στα πλαίσια της επέμβασης στο σώμα τους και χτυπάει βέβαια το σύστημα κάθε φορά που περνάνε και ενοχλούνται πάρα πολύ. Επομένως, επί της αρχής υπάρχει η υποδομή, ο μηχανισμός για να αποφύγουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Υπάρχει υποδομή προκειμένου να αποφύγουμε την πλήρη σωματική απεικόνωση, απεικόνηση και νομίζω ότι σε αυτό ακριβώς θα πρέπει να επιμείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα, κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές στις υποδομές μας. Νομίζω ότι το αεροδρόμιο του Σίπολ στην Ολλανδία χρησιμοποιεί κάτι τέτοιο. Ολοκληρώντας να πω ότι αναφερθήκατε στο ζήτημα του passenger profiling, του προφίλ του επιβάτη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τα κράτη-μέλη και νομίζω ότι θα πρέπει να ενισχυθούν τα μέτρα κατά της τρομοκρατίας καθώς επίσης και ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στα κράτη-μέλη γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να προχωρήσουμε σε όλα αυτά τα μέτρα και να μην υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Νομίζω ότι τα κράτη-μέλη και σε διεθνές επίπεδο θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταλλάσσουν τις πληροφορίες αυτές. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Ρικέ. Δύο λεπτά είναι ο χρόνος που έχετε. Ευχαριστώ. Ποιο είναι το πρώτο που θέλω να πω. Οι νέες τεχνολογίες απεικόνησης ε, ξεπερνά ιδιαίτερα αυτό το πρόβλημα που είναι για τα αεροδρόμια, έτσι. Αυτή η τεχνολογία θα επεκταθεί νομίζω σε όλο το σύστημα ελέγχου ασφαλείας, έτσι. Είναι το θέμα ιδιαίτερα ευρύ. Δεύτερη παρατήρηση τώρα. Υπάρχουν προβλήματα αρχής καθώς και ανάπτυξης ε, τεχνολογικής. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να σεβαστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, σεβασμός της αξιοπρέπειας, απόλυτα θα πρέπει να γίνει σεβαστό αυτό. Τώρα το πρόβλημα που έχει να κάνει με τη τεχνολογία δύσκολα θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο ενός κανονισμού. Τώρα η αποτελεσματικότητα εξαρτάται μέσα από την τεχνολογία που χρησιμοποιείται, τι παρατηρούμε, τα μικροκύματα, εντάξει μπορούν να βελτιωθούν αυτά ιδιαίτερα ε, και διάφορα άλλα συστήματα επίσης. Ε, τώρα το η αποτελεσματικότητα δεν ξέρω πώς θα ενταχθεί σε ένα ε, κανονισμό εκτός αν αφήσουμε ανοιχτή μια πορτούλα τώρα και το κόστος όφελος ε, αυτό δεν ξέρω αλλά υπάρχει μια πραγματική δυσκολία για να μπει στα πλαίσια ενός κανονισμού ε, να ενταχθεί σε ένα κανονισμό ενώ η αρχή δεν είναι δύσκολο Εντάξει, η αρχή αυτή για ένα ευρωπαϊκό κανονισμό είναι κάτι πολύ σημαντικό και ίσως καταλήξει σε μια ε, γενική χρησιμοποίηση και πέρα από τα αεροδρόμια. Η υποχρέωση αποτελέσματος είναι, αλλά όχι μέσω σε περίπτωση ασφαλείας και θα μπορούσε να αποτελέσει έτσι αντικείμενο ε, για κάτι το αναγκαστικό, υποχρεωτικό. Είναι κάτι που ξεπερνάει ιδιαίτερα αυτόν τον κανονισμό ο οποίος αναφέρεται. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριο Ρικέλε, πρόεδρος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να γνωρίζω αν η Αντιπρόεδρος Ρέντινγκ συμμετείχε στις συζητήσεις που γίναν και στις διαβουλεύσεις και αν συμφωνεί με την ακίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί δεν με ικανοποιεί ιδιαίτερα. Νομίζω ότι α, δεν ασχολείται όσο θα έπρεπε με το ζήτημα της αναλογικότητας όσον αφορά την ασφάλεια και όσον αφορά τη χρησιμοποίηση των ε, σαρωτών. Νομίζω ότι θα ήταν καλύτερα το κείμενο να προσπαθεί να ε, προλάβει αν θέλετε κάποια επικίνδυνα φαινόμενα. Πουθενά δεν βλέπω στο κείμενο αυτό ποιες ακριβώς είναι οι τεχνολογίες αυτές που θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν Πολύ συχνά στο παρελθόν χρησιμοποιούμε αναφορές σε λογισμικά τα οποία υποτίθεται ότι θα μας βοηθήσουν να αποφύγουμε κακή χρήση της υποδομής και πολλές φορές δεν λειτουργούν καν σωστά. Νομίζω ότι ο μόνος τρόπος για να αποφύγουμε την ε, αποθήκευση και μεταφορά των ε, πληροφοριών, θα έπρεπε να μην προβλέπετε κάτι τέτοιο στην ίδια τη μηχανή, να μην μπορεί να αποθηκεύει δηλαδή το ίδιο το μηχάνημα της πληροφορίας. Εσείς λέτε όμως ότι το μηχάνημα αυτό θα πρέπει να διατηρεί τις ε, πληροφορίες για να ελεγχθούν εκ των υστέρων. Άρα το μηχάνημα θα τι αποθηκεύει τελικά, θα τι κρατά τι πληροφορίε αυτέ. Αναφερθήκατε επίση σε νέα μηχανήματα που ε, χρησιμοποιούν νέε τεχνολογίε, τη τεχνολογία της αυτόματη, του αυτόματου εντοπισμού των απειλών. Αυτό που βλέπουμε όμω είναι ότι υπάρχουν πολλά εθνικά κέντρα έρευνα που λένε ότι οι μηχανισμοί αυτοί δεν είναι ακόμα πάρα πολύ ακριβεί. Όσον αφορά το opt-out, από τη μια, η έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής λέει ότι ο έλεγχος που γίνεται με τα χέρια είναι εξίσου αποτελεσματικός με τους σαρωτές, αλλά από την άλλη λέτε ότι ε, δεν προβλέπεται η δυνατότητα του ε, opt-out ή ότι δεν υπάρχει δυνατότητα χρησιμοποίησης του, της μίας ή της άλλης μεθόδου. Δεν, καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν να τα βάζετε και τα δύο ουσιαστικά μέσα στην ε, έκθεση αυτή. Σας ευχαριστούμε κυρία Λούτφορτ. Van Orden. Κύριε Πρόεδρε, μην ξεχνάμε γενικά ποιο είναι το όλο εγχείρημα εδώ πέρα. Θέλουμε να αποφύγουμε τις τρομοκρατικές πράξεις και θα πρέπει να βοηθήσουμε και τους νομοταγείς ταξιδιώτες να ταξιδεύουν ευχάριστα, άνετα και να περνάνε άντα μέσα από τα αεροδρόμια. Δεν φαίνεται ότι τα έχουμε αυτά τα δύο κατά νου. Οι τρομοκράτες πάντα θα ψάχνουν τον αδύναμο κρίκο. Συμφωνώ με την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε διάφορα επίπεδα και την ανάλυση που γίνεται για τον ανθρώπινο παράγοντα, human factor analysis. Επίσης, πρέπει να δούμε όλους αυτούς οι οποίοι έχουν πρόσβαση στα αεροδρόμια και μπορούν να αποτελέσουν τον αδύναμο κρίκο. Θέλουμε καλά συστήματα εποπτείας, αυτό δεν υπάρχει πάντα νομίζω ότι θα πρέπει ενδεχομένω να έχουμε και ένα σύστημα ασφαλούς επιβάτη, αν θέλετε. Προσπαθώ και εγώ να δω ακριβώ ποια είναι η χρησιμότητα των ε, σαρωτών. Νομίζω ότι εφόσον χρησιμοποιούμε σαρωτέ θα πρέπει η τεχνολογία που χρησιμοποιείται να είναι εύχρηστη. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν ανησυχίε όσον αφορά την υγεία και άλλου τομεί. Και Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι νομίζω ότι αφαίρεντα αντιτίθενται αυτή τη στιγμή στην εισαγωγή τη νέα τεχνολογία. Αν γίνει μια τρομοκρατική επίθεση αύριο μεθαύριο, νομίζω ότι όλοι αυτοί θα σοπάσουν και θα συμφωνήσουν με την χρησιμοποίηση τη νέα αυτή τεχνολογία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι ορισμένα αεροδρόμια δεν τηρούν καλά πρότυπα, δεν έχουν καθόλου πρότυπα. Ποιο είναι ο ρόλο όμω τη ε, Διεθνή Αρχή Πολιτική Αεροπορία. Νομίζω ότι δεν πρόκειται μόνο για ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Υπάρχουν σαφώ κάποια αεροδρόμια στην Ευρώπη που πιστερούν, αλλά υπάρχουν και αεροδρόμια που πιστερούν ακόμα περισσότερα εκτό Ευρώπη. Ο κύριο Δεγκράντε Πρεσίδεντη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για την Επιτροπή να πω είναι ότι στην συζήτηση για το 2008 τότε όλοι ασκήσαμε κριτική, έτσι. Στην περίπτωση αυτή πιστεύω, το λέω, ότι εκπλήρωσε την αποστολή της, ε, του Οκτωβρίου του 2008 είναι σοβαρή, δεν είναι δογματική αυτή η έκθεση. Ξεκινάει μια συζήτηση για το Κοινοβούλιο και για το Συμβούλιο και θα πρέπει να δούμε για την εκπλήρωση αυτή της εντολής σε σχέση με θέμα τα που λέγαμε ότι έπρεπε να αντιμετωπίσουμε. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει μια λύση για τα πάντα, αλλά ξεκινάει ένα δρόμο. Εδώ θα πρέπει και στην Επιτροπή επίσης Δημοσιολευθεριών να ξεκινήσει και εδώ και όλα αυτά τίθενται νομίζω σε καλή βάση από την Επιτροπή ορισμένα συμπεράσματα που εμφανίζονται στην έκθεση, σοβαρά συμπεράσματα, έστω και αν δεν είναι πλήρως αποτελεσματικά πλήρη. Εδώ έτσι με νομικό τρόπο θα μπορούσαμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις ε, προδιαγραφές. Όλα αυτά που αναφέρονται είναι σοβαρά και αυστηρά και θα πρέπει με την τεχνολογία να εξασφαλίσουμε και την υγεία και το σεβασμό των βασικών θεμελιωδών δικαιωμάτων εσωτόμου και αυτό είναι πολύ σοβαρό συμπέρασμα. Οποιαδήποτε τεχνολογία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ότι θα πρέπει να χρησιμοποιεί ερμόνηση ε, και να υπάρχει και ένα εναλλακτικό σύστημα για τα ευαίσθητα σε ορισμένε ε, εξετάσει ε, άτομα και αυτό είναι σοβαρό. Και επίση θα πρέπει να δούμε τι γίνεται πριν από τη χρησιμοποίηση αυτών των τεχνολογιών. Θα πρέπει όλα αυτά να μιληθούν Νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρό πλευρά Επιτροπή. Η Επιτροπή νομίζω ότι εκπλήρωσε την αποστολή τη. Είναι σοβαρή αυτή η συζήτηση και κάθε μια από αυτέ τι υποθέσει τι αναλύουμε και εδώ και στην Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών. Όπω είπε κάποιο Έγκλο συνάδελφο, ε, δεν ξέρουμε πώ μπορεί να σταματήσει ο, η τρομοκρατία δεν νομίζω σταματάει. Δεν πρέπει να ησυχάσουμε λοιπόν. Ε, θα πρέπει να δούμε, να προχωρήσουμε, να προσπαθήσουμε χωρίς καμία πάυση, χωρίς καμία διακοπή σε όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με το σύνολο της Ευρωπαϊκής Κοινωνίας. ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Λάιχτριντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με πολλά από αυτά τα οποία ακούστηκαν. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση και δύο παρατηρήσεις. Το ερώτημα. Δεν αντιλαμβάνομαι πώς μπορούμε να έχουμε ένα σύστημα το οποίο δεν θα είναι ενιαίο στην Ευρώπη, γιατί λέτε όσοι θέλουν τελικά μπορούν να το κάνουν και να έχουμε μετά ένα σύστημα One Stop Security. Μου φαίνεται αντιφαντικό γιατί αν κάποιος ε, απλά διαλέξει άλλο αεροδρόμιο μπορεί να μπει χωρίς ε, σαρωτή. Μετά να αναφέρω δύο πράγματα. Είπατε πως βλέπετε την πολιτική ευαισθησία του ζητήματος. Αλλά δεν νομίζω εάν όντως κάνετε αυτά τα οποία θέλετε να κάνετε ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Εάν ακούσουμε δηλαδή Συμβούλιο και Κοινοβούλιο νομίζω πως δεν επαρκεί επιτροπολογία για αυτή τη διαδικασία. Εάν αποφασίσουμε οι ίδιοι ε, πως είμαστε δυσαρεστημένοι με κάποια πράγματα τα οποία προτείνει η Κομισιόν. Δεύτερον, πρέπει να βρεθεί και μια λύση για τη χρηματοδότηση. Και γνωρίζουμε όλοι πως ε, το μπλοκάρισμα της χρηματοδότησης αυτή τη στιγμή οφείλεται στο Συμβούλιο. Και έχω συζητήσει με πολλούς ε, συναδέλφους και κάποιοι θεωρούν πως αυτά τα πράγματα πρέπει να λυθούν παράλληλα. Και αν το Συμβούλιο δεν είναι σε θέση να δει το ζήτημα της χρηματοδότησης και να βρει μια και λύση μαζί μας, τότε το Κοινοβούλιο θα μπορούσε νομίζω να φέρει και αυτό τις αντιρρήσεις του σε αυτός. Ευχαριστώ κύριε Στέρξ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος ονόματος του συναδελφού Ρούτζας, ο οποίος δεν είναι εδώ βρίσκεται σε κάποια επίσκεψη. Ο κύριος Ούτζας λοιπόν θα καταθέσει μια γραπτή ερώτηση για αυτό το ζήτημα και αναμένει μια γρήγορη απάντηση. Ευχαριστώ. Thank you, short and sweet. Mr. Van Dalen. Έτσι σύντομα και ωραία, κύριε Φαντάλεν. Κύριε Πρόεδρε, έχω ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα στον κύριο Ρούτε. Κύριε ρίτε υποθέτω πως ένας τρομοκράτης αναζητεί βεβαίως πάντα τον πιο αδύναμο κρίκο της αλυσίδας, δηλαδή στην ευρωπαϊκή αεροπορία. Εάν ξεκινήσουμε με αυτό το ερώτημα, το ερώτημα είναι, αντιλαμβάνομαι από το έγγραφο πως λέτε πως τα κράτη-μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν έναν τέτοιο σαρωτή. Αν σκεφτεί δηλαδή πού θα μπει πιο εύκολα ο τρομοκράτης, θα μπει από τα μέρη εκείνα τα οποία δεν χρησιμοποιείται ο σαρωτής. Πέραν βεβαίως των προφίλ και της ανθρώπινης ανάλυσης. Γιατί λοιπόν δεν γίνεται η υποχρεωτική ή χρήση στα αεροδρόμια που έχουμε πάνω από ένα εκατομμύριο επιβάτες. Και μάλιστα ε, συγκεκριμένα τον ε, τύπο εκείνος ερωτών που δεν, δεν προκαλεί επιπλέον ε, πρόβλημα και βάρος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε εκπρόσωπε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε για το ζήτημα της ασφάλειας, γιατί ακριβώς αυτό περιμένουν από εμά και οι Ευρωπαίοι πολίτες. Ανταλλάσσουμε αυτή τη στιγμή απόψεις για ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με την ασφάλεια. Μιλάμε πιο συγκεκριμένα για τους σαρωτές σώματος. Πρωτού όμως προχωρήσουμε παραπέρα στη συζήτηση, νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε κάποια συγκεκριμένα δεδομένα. Την προηγούμενη εβδομάδα ένας πολίτης της Ρουμανίας πήγε, πήρε το αεροπλάνο για να πάει από την Βιέννη στο Λονδίνο. Στη συνέχεια, ένας ε, Ιταλός δημοσιογράφος έδειξε ότι μεταξύ του, ε, της μία, μία και τριών το πρωί στο Φιουμιτσίνο υπάρχουν, υπήρχε ένας συγκεκριμένο αριθμός ε, μεγάλος επιβατών που δεν περνούσε καθόλου από έλεγχο. Επίσης, σε άλλο αεροδρόμιο βρέθηκε κάποιος ο οποίος έγραψε με γκράφιτι πάνω σε ένα αεροπλάνο και κανείς δεν τον σταμάτησε. Για ποιο λόγο λοιπόν έχουμε τόσο ακριβά μηχανήματα ασφάλειας όταν βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή, οποιαδήποτε στιγμή μπορεί κανείς να μπει σε ένα αεροδρόμιο, να επιδείξει το φράκτη και να κάνουν τι με στο αεροδρόμιο αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε για τους ε, σαρωτέ σώματος αυτή τη στιγμή, αλλά το ερώτημα το οποίο θα ήθελα να θέσω είναι ότι ε, μπορούν οι σαρωτέ αυτοί να πετύχουν ένα ε, ίσο επίπεδο ασφάλειας σε όλες τις χώρες. Πριν από λίγο καιρό ήμουνα στο αεροδρόμιο των Βρυξελών και Παρατηρώντα το αεροδρόμιο, συνειδητοποίησα ότι υπήρχαν τουλάχιστον δύο τρόποι που θα μπορούσε κανεί να περάσει από τον έλεγχο, μεταφέροντα ακόμα και μία βόμβα. Οι Ιταλοί μιλάνε ακόμα και για σερωτέ σώματο αυτή τη στιγμή θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στα τρένα. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουν με τα αεροδρόμια καλύτερα. Uh, Ο κύριος Μπράντμπορν θα ήθελα να αφαιρθώ σε ένα πράγμα πρωτού περάσω σε δύο βασικές αρχέ θα μπορούσε η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πει εδώ πέρα ότι μιλάμε για σαρωτές σώματος, για σαρωτές που καλύπτουν όλο το σώμα. Αυτό. Τώρα. Πριν από λίγο είπαμε αν θα πρέπει οι μηχανές αυτές να χρησιμοποιούνται με θελούσιο τρόπο ή αν θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίησή τους. Ήμουνα στην Οτάβα τον προηγούμενο μήνα και μίλησα στην ε, Καναδέζικη Υπηρεσία για τις Μεταφορές και εκεί πέρα χρησιμοποιούν μία άλλη μέθοδο. Για ποιο λόγο να μην κάνουμε κι εμείς το ίδιο πράγμα στην Ευρώπη. Γιατί βλέπετε ότι κανείς δεν αντιτίθεται στο στη μέθοδο αυτή ούτε στον Καναδά ούτε στι Ηνωμένε Πολιτείε, που προεγραφές ασφάλεια είναι πάρα πολύ υψηλές. Χρησιμοποιούν σε κάποια αεροδρόμια μόνο το σύστημα ελέγχου με τα χέρια. Επίσης, οι σαρωτέ αυτοί άρχισαν να χρησιμοποιούνται σαν αντίδραση σε κάτι το οποίο δεν θα μπορούσαμε καν να εντοπίσουμε στο παρελθόν. Δηλαδή αναφέρομαι στα υγρά εκείνα τα οποία θα χρησιμοποιούσε επιβάτη στην πτήση από το Άμστερνταμ στο Ντιτρόιτ. Νομίζω ότι ούτε και ένα σαρωτή σώματο δεν θα έχει καταφέρει καν να εντοπίσει τα υγρά αυτά. Για ποιο λόγο λοιπόν οι συγκεκριμένοι σαρωτέ ε, σώματο, με συγχωρείτε, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Υπάρχουν και άλλοι σαρωτέ οι οποίοι χρησιμοποιούν την οσμή, χρησιμοποιούν υπερήθρια ακτινοβολία, δεν χρησιμοποιούν το σύστημα τη απεικόνηση, δεν έχουν καθόλου καθόλου Για ποιο λόγο να μην συμπεριλάβουμε και τα μηχανήματα αυτά στι που προβλέπει το έγγραφο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και επ' αυτού, κύριε, κύριε Πρόεδρε, η χρησιμοποίηση των ακτίνων Χ ή χρησιμοποίηση ακτίνων Χ με οπισθοσκέδαση νομίζω ότι δεν θα πρέπει να προβλέπεται καθόλου. Θα πρέπει να απαγορευτούν γιατί ακριβώ υπάρχουν κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία. Κυρία Γιάλα <clears throat> ναι. Σέντερ. Προχωράω εδώ. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο και αυτό για να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε την ολυπορία. Δεν ε, θα πρέπει να προκαλεί κάτι το αρνητικό για αυτούς τους αρωτές. Εδώ ρωτάω τον συνάδελφο τι θα γίνει εάν απορρίψουμε την πρόταση της Επιτροπής. Ε, κάτι παρόμοιο τι επίπτωση θα είχε και τι θα γίνει και ε, βέβαια με ιδιαίτερα επιχειρήματα που έχουν να κάνουν με την υγεία είτε με την ιδιωτική σφαίρα ζωής, τι θα γίνει τότε με τα κράτη-μέλη, πώς όλα αυτά θα επηρέαζαν τα κράτη-μέλη. Συμφωνώ με την αποτελεσματικότητα και γι' αυτό το λόγο να αποφύγουμε να ενοχλούμε τους ε, ε, επιβάτες, ε, αλλά για την Επιτροπή, εντάξει, για τα 20 λεπτά, Εντάξει, όταν κάναμε την παρουσίαση είχαμε διαφερθεί όλοι μας. Αυτή ήταν από τα σημαντικά που ρωτούσαμε Μήπως ε, δεν ε, θα μπορούσε να μειωθεί ο χρόνος που περνάνε από εκεί οι επιβάτες. Λέμε ότι θα έχουμε κρίσεις, ε, κρίσεις θα έχουμε μια αύξηση στο μέλλον. Εντάξει μιλάει για αυτό το ενδεχόμενο και για την υγεία, οι ακτίνες χ δεν ξέρω τι θα γίνει με την τεχνολογία, αν χρησιμοποιηθεί αυτή η τεχνολογία. Είναι από εκείνες που χρησιμοποιούνται σήμερα. Ε, μιλάμε για χαμηλές τιμές. Ε, κάποια στιγμή λέει όμως ότι μια κάποια αύξηση, γιατί σιγά σιγά με μια, ε, με μια συγκέντρωση θα μπορούσαν να ξεπεραστούν οι ετήσιες τιμές έκθεσης. Έτσι, γιατί αναφέρεται ότι εντάξει στο μέλλον θα υπάρξει μια νέα τεχνολογία. Κάτι ακόμα θα ήθελα να σας ρωτήσω εδώ, εάν ε, με τον ε, Ευρωπαίο ε, ελεγκτή της υγείας του πολίτη αν υπήρξε μια διαβούλευση. Τι καλ. Ναι. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα επαναλάβω εγώ ότι είπαν ήδη οι συνάδελφοι. Τον κύριο Βόλτον θα ήθελα να ευχαριστήσω για την παρουσίαση εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που πολύ σοβαρά αναλύει όλα αυτά για πώς επηρεάζεται η υγεία και την αποτελεσματικότητα αυτών των ε, μεθόδων ε, και τι γίνεται, πώς θα αποφύγουμε, πώς θα σεβαστούμε τα θεμελιώδη δικαιώματα και όλα αυτά έχουν σημαντικά και στην τεχνολογία και στην όλη διαδικασία. Τώρα για τον τρόπο χρησιμοποίηση αυτών των σαρωτών και την προστασία των προσωπικών δεδομένων ε, πρέπει να προχωράει κανείς πεντακάθαρα και να μην γίνεται μια οποιαδήποτε παραβίαση της ιδιωτικής σφαίρας ζωής. Και κάτι να σας ρωτήσω, εκεί όπου χρησιμοποιείται αυτός ο σαρωτής, εντάξει σε θελούσια βάση, πέστε μου κάτι οι επιβάτες μπόρεσαν να αντιδράσουν αν ήθελαν τη στιγμή που περνούσαν τα, το σαρωτή αυτό. Κούρτ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, δύο ερωτήσεις. Από ό,τι ακούω, φαίνεται πως θα έρθει ούτως ή άλλως ο σαρωτής αυτός Απλά θα ήθελα να γνωρίζω πώς συμπεριφέρεται το σύστημα αυτό σχέση με άλλες ε, μεθόδους ε, και το τι λένε οι υπηρεσίες ασφάλειας. Δεύτερον, στην σημερινή ανακοίνωση η Κομισιόν λέει στην ε, παράγραφο 89 πως πρέπει να ληφθεί μια απόφαση για ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για τη χρήση των σαρωτών και, μετά, και θα ακολουθήσει μία αξιολόγηση αντικτύπου. Εάν δεν γίνει κάτι τέτοιο και πάμε στα εφαρμοστικά μέτρα, θα γίνει ούτως ή άλλως μια αξιολόγηση αντικτύπου. Για... Θα έχουμε μετά λόγο ως ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με συγχωρείτε, στην περίπτωση που πάει στην ε, διαδικασία της Επιτροπολογίας. Η κυρία Γουίλς, ναι, ευχαριστώ όπως είπατε δεν ε, έχει γίνει καμία έρευνα για την ε, αναλογικότητα και σε σχέση με τις υπάρχουσες ε, τεχνολογίες. Οπότε είναι νομίζω και θέμα αξιοπρέπειας. Ποιες εικόνες δημιουργούνται και που αποθηκεύονται και είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που, και οι βουλευτές που το κάνουν αυτό, πετάνε για τη δουλειά τους. Επίσης τι γίνεται με ανάπηρους εγγύους παιδιά και την ακτινοβολία αυτή, την αποθήκευση των δεδομένων, ποιος αποθηκεύει τα δεδομένα, πώς χρησιμοποιούνται, πάνε σε ευρωπαϊκό, σε εθνικό δίκτυο και όταν μιλάμε για αποθήκευση δεδομένων πάντα υπάρχουν άνθρωποι που θα τα χρησιμοποιήσουν λάθος και με εγκληματικό τρόπο. Δεν θέλω οι εικόνες μου να καταλήξουν και να απολούνται κάπου σε ανθρώπους που θέλουν να βγάλουν ε, λεφτά. Υπάρχουν λοιπόν πολλές ε, ερωτήσεις ε, και εγώ επί της αρχής είμαι κατά του να εισαχθεί αυτό το σύστημα έτσι όπως προτείνεται. Ευχαριστώ κύριε Βίλς, κύριε Ρόιτε πριν απαντήσετε τις ερωτήσεις να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την πειθαρχία τους. Ξέρω πως στην Ισπανία μου λέγατε πως διευθύνεται την Επιτροπή πρόσος και το θεώρησα κομπλιμέντο. Ελπίζω όμως να αντιλαμβάνεστε πως ε, όταν έχουμε ένα τέτοιο κατάλογο ομιλητών πρέπει να είμαστε πειθαρχημένοι και σας ευχαριστώ για τη συνεργασία σας σήμερα και την πειθαρχία που επιδείξατε. Για να μιλήσουν όλοι και να μπορέσει να απαντήσει και ο κύριος Ρόιτερ. Ε, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να απαντήσω σε ερωτήσεις σας, ώστε να το γρηγορότερα. Θα ξεκινήσω μετά όσο είπε ο κύριος Γκρός. Ας πάμε ένα βήμα πίσω και δούμε τα πράγματα με κάποια απόσταση. Τι θέλουμε ακριβώς να πετύχουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μάλλον έχουμε ένα κανονισμό που λέει ακριβώς τι είδους μέτρα μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ελεγκτές στα αεροδρόμια προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξει στο αεροσκάφος καμία βόμβα ή κανένα όπλο. Στον κανονισμό λοιπόν αυτό έχουμε διαφορετικές μεθόδους που προβλέπονται. Έλεγχος με τα χέρια, οι πύλες ανείχνευσης μεταλλικών αντικειμένων, σκύλοι οι οποίοι μπορούν να εντοπίσουν εκρηκτικές ουσίες, μηχανήματα χειρός τα οποία χρησιμοποιούνται για την ανείχνευση μεταλλικών αντικειμένων και να πρόκειται σε κάθε κράτος μέλος να αποφασίσει ποια θα χρησιμοποιήσει και πώς θα τα συνδυάσει μεταξύ τους. Όταν λοιπόν ήρθαμε σε επαφή μαζί σας την πρώτη φορά, αρχίσαμε να μιλάμε στη συνέχεια για τους ε, σαρωτές ε, σώματος ως ένα επιπλέον μηχανισμό ανείχνευσης. Έτσι έχουν τα πράγματα, αυτή είναι η συζήτηση που κάνουμε και έχετε σαφώς το δικαίωμα εσείς αρνηση όσον αφορά την ε, εναλλακτική αυτή λύση που που σας προτείνουμε. Τώρα έχουμε και τους εφαρμοστικούς κανόνες που θα πρέπει και αυτοί να εγκριθούν μέσω της διαδικασίας της επιτροπολογίας. Και νομίζω ότι και εξ ονόματος του Αντιπρόεδρου Κάλλας μπορώ να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε ποιοι θα είναι οι εφαρμοστικοί κανόνες οι οποίοι θα συνοδεύσουν την νομοθεσία για τους αρωτές σώματος. Εφαρμοστικοί κανόνες στους οποίους θα αναφέρεται με κάθε λεπτομέρεια ποια υποδομή θα χρησιμοποιηθεί, ποια τεχνολογία θα χρησιμοποιηθεί, ποιοι κανόνες θα πρέπει να εφαρμόζονται όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, όσον αφορά το να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχει καμία εικόνα η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με άλλο τρόπο. Αυτοί λοιπόν οι εφαρμοστικοί κανόνες θα αποτελούν μια ξεχωριστή δέσμη μέτρων, γιατί δεν μπορείτε εσείς απλώς να πείτε ναι στην αρχική πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει να δείτε σφαιρικά την όλη νομοθεσία συμπεριλαμβανομένων των εφαρμοστικών κανονισμών. Θέλουμε λοιπόν εμείς να έχουμε μια πάρα πολύ καλή σύντηση μαζί σας για το πώς θα πρέπει να διαμορφωθεί αυτή η δέσμη μέτρων προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα επιπλέον νομοθετικό μέσο εφόσον αξίζει να δημιουργηθεί σαφώς ένα επιπλέον νομοθετικό μέσο το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα κράτη-μέλη. Ο Μάθιου Γκρος το είπε πολύ καλά ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε ένα επίπεδο ασφάλεια 100%. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα απόλυτο επίπεδο ασφάλεια. Και θα πρέπει να έχουμε κάποιου ε, ευρωπαϊκού κανόνε όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όσον αφορά την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, όσον αφορά την προστασία τη υγεία. Πρέπει όμως να εξασφαλίσουμε ότι ε, Μάλλον θα πρέπει να δούμε ότι αυτή τη στιγμή ισχύει και άλλη νομοθεσία. Υπάρχει μια υφιστάμενη νομοθεσία όσον αφορά τα υγρά, με την οποία έχετε συμφωνήσει και εσείς βέβαια, και εγκρίναμε την νομοθεσία αυτή προκειμένου να σταματήσουμε τον έλεγχο που, γινόταν για τις, που γίνεται ακόμα για τα υγρά, προκειμένου να σταματήσει ο έλεγχος αυτός. υπάρχει μια νέα υποδομή, μια νέα τεχνολογία που θα αρχίσει να ισχύει από τον Απρίλιο και που θα δίνει τη δυνατότητα κατά αυτόν τον τρόπο στους επιβάτες να μπορούν πιο εύκολα να μεταφέρουν ε, εμπορεύματα που έχουν αγοράσει στα duty free και στη συνέχεια θα έχουμε μία νέα μέθοδο που θα μας επιτρέπει να μην χρειάζεται πλέον οι επιβάτες να κουβαλάνε αυτές τις φραγισμένες σακούλες όσον αφορά τα προϊόντα τα οποία έχουν αγοράσει. Θεωρώ λοιπόν ότι η χρησιμοποίηση αυτών των σαρωτών σώματος θα μας βοηθήσει να σταματήσουμε πλέον την χρησιμοποίηση αυτών των ανοιχνευτών μετάλλων, αυτής της πύλης ανοίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων που έχουμε τώρα στα αεροδρόμια. Δεν θα έχουμε πλέον αυτή την πύλη ανοίχνευσης, δεν θα έχουμε αυτά τα 20 δευτερόλεπτα, δεν θα έχουμε την ακνοβολία που χρησιμοποιούν τα μηχανήματα αυτά θα έχουμε μηχανήματα τα οποία θα μπορούν να ελέγχουν και τα μεταλλικά αντικείμενα αλλά παράλληλα και τις υγρές ουσίες. Επομένως, τα επόμενα χρόνια πραγματικά πιστεύω ότι με τη νέα αυτή τεχνολογία τα ταξίδια θα γίνουν πιο εύκολα. Έτσι βλέπω εγώ τα πράγματα. Πρέπει αφενός να δούμε τον ίδιο τον επιβάτη και ξεχωριστά βέβαια και τα αντικείμενα αυτά τα οποία ο επιβάτης αυτός μεταφέρει μαζί του. Τώρα, πώς τα νέα αυτά στοιχεία επηρεάζουν τα αεροδρόμια. Νομίζω ότι αυτό θα μας το πει και η μελέτη αντικτύπου, εφόσον βέβαια γίνει και όταν ολοκληρωθεί. την ίδια στιγμή με συμφωνίες που έχουμε με τρίτες χώρες θα είμαστε ενδεχομένως σε θέση να έχουμε μία και, μία και μόνη θηρίδα ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συζητάμε αυτή τη στιγμή με τις Ηνωμένε Πολιτείες, δηλαδή μια πτήση που φεύγει από τις Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη συνέχεια ελέγχεται πάλι στην Ευρώπη εφόσον η πτήση αυτή συνεχίσει για μία άλλη χώρα. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ισότιμο επίπεδο ασφάλειας όπου θα αρκεί ένας και μόνο έλεγχος. Κατά αυτόν τον τρόπο θα διευκολύνουμε περισσότερο και τους ίδιους επιβάτες. Ο κύριος Τσιζάντα αναφέρθηκε σε διάφορα αεροδρόμια όπου η ασφάλεια δεν είναι πολύ καλή ακόμα, τα επίπεδα ασφάλειας εστερούν. Εμείς γνωρίζουμε την κατάσταση αυτή και μάλιστα κάνουμε και τους απαραίτητους ελέγχους προκειμένου να εντοπίσουμε ότι υπάρχει το επιθυμητό επίπεδο ασφάλειας. Αυτό γίνεται επιπλέον με όλα τα άλλα τα οποία κάνουμε για να εξασφαλίσουμε ένα καλό επίπεδο ασφάλειας. Κύριε Ελκαντράουι, θέστε το σωστό ερώτημα. Τι θα γίνει μετά την περίοδο αυτή των 13 μηνών. Τους πρώτους 30 μήνες μάλλον τι γίνεται. Κοιτάξτε. Έχουμε διαφορετικούς κανόνες αυτή τη στιγμή για τη χρησιμοποίηση των μηχανημάτων αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά την πάροδο των 30 αυτών μηνών φοβάμαι ότι οι κανόνες θα γίνουν πιο αυστηροί θα έχουμε έναν πιο αυστηρό κανόνα, σύμφωνα με τον οποίο θα πρέπει να γίνει μια πολύπλοκη ανάλυση κόστους-οφέλους, να δούμε αν τελικά δικαιολογείται η εφαρμογή του κανονισμού αυτού. Πάντως τον κανονισμό 300 προβλέπεται η δυνατότητα να έχουμε κάποιους κοινού κανόνες που θα εγγυώνται παράλληλα και τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προστασία της υγείας. Ο κ. Ελκαντράνου, καθώς επίσης και κάποιοι άλλοι βουλευτές, αναφέρθηκαν στο ζήτημα του κόστους. Όντως αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μια συζήτηση ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για το αν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν επιπλέον οι πιο αυστηρά μέτρα ασφαλείας και αν θα πρέπει το κόστος τελικά να το ο φορολογούμενος ή τα αεροδρόμια. Δεν θα ήθελα να προεξοφλήσω αυτή τη στιγμή την έκβαση της συζήτησης. Βλέπω πάντως τι θέλετε να πείτε. Καταλαβαίνω ποιο είναι το σχόλιο σας. Όταν κάναμε άλλωστε την πρόταση εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πηγαίναμε κι εμείς προς την κατεύθυνση αυτή την οποία εσείς περιγράψατε. Δεν θα είμαι σε θέση να απαντήσω φοβάμαι σε όλες τις ερωτήσεις Το ζήτημα του κόστους πιστεύω και εγώ ότι είναι σημαντικό, θα πρέπει να μας απασχολήσει, αλλά γενικά αυτό που θα έλεγα είναι ότι αν είναι να τροποποιηθεί τελικά ο κανονισμός, αν προσθέσουμε στον κανονισμό και τους αρωτές ασφάλειας ή σαρωτές σώματος όπως θέλετε και αν μπουν και αυτοί οι αρωτές στον κατάλογο των εναλλακτικών μέσων ελέγχου της ασφάλειας, τότε είναι σαφές για μένα ότι δεν θα είναι υποχρεωτική η χρήση τους, όπως δεν είναι υποχρεωτική και η χρήση α, σκύλων. Δεν θα είναι υποχρεωτικό δηλαδή να υπάρχει σε κάθε αεροδρόμιο και να ρωτήσει σώματος. Κατά πάση πιθανότητα όμως τα μεγαλύτερα αεροδρόμια θα πρέπει να εξοπλιστούν και θα χρησιμοποιήσουν τους ερωτές αυτούς γιατί είναι θετική τόσο για την ασφάλεια όσο και για το ζήτημα του κόστους. Και τα άλλα αεροδρόμια ενδεχομένως να συνδυάσουν με πιο αυστηρό τρόπο τους, τις άλλες μεθόδους ελέγχου. Είναι πιστεύω σαφές και το είπαν και πολλοί βουλευτές, η κυρία Φώστερ μεταξύ άλλων, στην αρχή, ότι Πρέπει να έχουμε μία κοινή προσέγγιση όσον αφορά την τρομοκρατία, την πάταξη της τρομοκρατίας. Γίνονται πολλές ε, διεργασίες προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι λαμβάνουμε υπόψη την δουλειά που κάνουν διάφοροι συνάδελφοι που ασχολούνται με το ζήτημα της εσωτερικής πολιτικής των εσωτερικών θεμάτων και σας διαβεβαιώ ότι την έκθεση αυτή, κυρία Λάτφορ, λέω και σε εσά, ότι συζητήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Κολέγιο των Επιτρόπων, και το σύνολο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποστηρίζει την έκθεση αυτή. Επίσης είναι σαφές ότι ε, υποστηρίζουν την ε, έκθεση αυτή γιατί έχει ξεκινήσει ήδη μία συζήτηση για πολλά από τα ζητήματα τα οποία θέτει η έκθεση αυτή. Τώρα όσον αφορά το διεθνές επίπεδο, ναι κύριε Βανόρντεν, όντως είναι σαφές ότι η ασφάλεια είναι διεθνές ζήτημα και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και στα πλαίσια του ΙΚΑΟ, αλλά στην πράξη αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπάρχουν πολλά κράτη στον κόσμο τα οποία ασκούν πίεση προκειμένου να σημειώσουμε πρόοδο στον τομέα της ασφάλειας. Αλλά παράλληλα υπάρχει και το γενικότερο ζήτημα της τρομοκρατικής απειλής που θα μπορούσε να έρθει από χώρες οι οποίες ε, δεν χρησιμοποιούν τόσο πολύπλοκα συστήματα σαν αυτά τα οποία χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ή ο Καναδάς ή οι Ηνωμένε Πολιτείε. Και γι' αυτό το λόγο στο πρόγραμμα εργασίας μας προβλέπεται μία ανακοίνωση στα τέλη του έτους που θα έχει να κάνει ακριβώς με το ζήτημα της ασφάλειας της ενέργειας κυκλοφορίας, ιδίως και τις πτήσεις από τις τρίτες χώρες, τις χώρες αυτές που υστερούν. Το ζήτημα αυτό θα απασχολήσει άλλωστε και τον ΙΚΑΟ σε μια συνδιάσκεψη που θα γίνει τον Σεπτέμβριο. Κύριε Μπράτμπορν, αναφερθήκατε στο παράδειγμα του Καναδά. Θέλω να είμαι απόλυτα σαφής. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο σας λέμε είναι το ακόλουθο ενδεχομένως να πρέπει να συμπεριλάβουμε τους αρωτές σώματος, σαρωτές ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ως έναν επιπλέον τρόπο ελέγχου. Το ζήτημα του τι θα γίνει αφότου εισαχθεί η νέα αυτή τεχνολογία σε ένα αεροδρόμιο. Τι θα γίνει δηλαδή με τις εγγύους, με τα άτομα ειδικέ ανάγκες, με τους ανθρώπους που αρνούνται να περάσουν από το μηχανισμό αυτό. Το ζήτημα αυτό δεν το έχουμε αναλύσει ακόμα. Θα πρέπει να το συζητήσουμε με εσά και θα πρέπει να αποτελέσει Ζήτημα το οποίο θα διευθετηθεί με τους εφαρμοστικούς κανόνες και βασιζόμαστε και σε εσά προκειμένου να, να καταφέρετε να μας βρείτε, αν θέλετε, το σωστό πλαίσιο το οποίο θα μας βοηθήσει να πετύχουμε την κατάλληλη ισορροπία, δηλαδή να μην έχουμε παραθυράκια στομοθεσία νομοθεσία για τους τρομοκράτες, αλλά από την άλλη να καταφέρνουμε επίσης να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις ανησυχίες που έχουν ακουστεί για την ανθρώπινη υγεία ή για την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Νομίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι απάντησα σχεδόν με γενικό πάντως τρόπο στις ε, ερωτήσεις. Αν υπάρχει τώρα κάποιος που πιστεύει ότι δεν απάντησα στην ε, ερώτησή τους, παρακαλώ πολύ κάντε μου σήμα και θα επανέλθω. Ευχαριστώ. Δεν θέλω τώρα να σηκώσετε όλοι τα χέρια σας για να ξεκινήσει η συζήτηση. Επί της διαδικασίας να είναι επί της διαδικασίας αν έχετε κάτι να πείτε και όχι ότι σας έρθει. Θα είμαι πολύ αυστηρός. Κύριε Λατφόρτ λοιπόν. Ναι κύριε Πρόεδρε. Ναι. Επί της διαδικασίας. Λέει ο κύριος Ρόιτε πως ξεκινά μια συζήτηση. Δεν έχετε προσέξει πως μένεται η συζήτηση τους τελευταίους 18 μήνες στον τύπο. Ελπίζω να, ελπίζω να κλείσει η Κομισιόν τη συζήτηση, να κάνει συστάσεις όπως αυτή η πράσινη βίβλος. Πώς ξεκινάτε τώρα την συζήτηση. Κυρία Λάτφορντ, λέει ο Πρόεδρος. Είστε και από την Βουλή των Λόρδων. Ξέρετε πως αυτό δεν ήταν επί της διαδικασίας, ήταν, ήταν σχόλιο. Ναι, ε, έτσι κάνουμε για να μπορέσουμε να μιλήσουμε. Λοιπόν. Τέλος, η κυρία Φώστερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένα θέμα θα ήθελα να αναφέρω το κύριο για το μέγεθος των αεροδρομίων. Είναι λάθος. Εάν είναι να έχουμε κανόνες για τους αρωτές πρέπει να είναι γενικοί. Γιατί να πάμε σε κάποιον και να του πούμε σε αυτό ναι, σε αυτό το αεροδρόμιο όχι. Είναι βλακώδες. Και τέλος για τον ε, εξοπλισμό. Νομίζω θα είναι προς το συμφέρον της Κομισιόν να χρησιμοποιήσει εξοπλισμό που δεν θα έχει προβλήματα και με την απεικόνηση και με την υγεία. Είναι εφικτό. Πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί σε αυτό, εάν θέμε να κινηθούμε. Κυρία Μποσκούρτ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι σαφές για μένα το τι σκοπεύει να κάνει η Κομισιόν. Θα έρθει νομοθεσία, θα περάσουμε σε εφαρμοστικές διατάξεις. Θέλω να το πω αυτό. Και δεύτερον, έφυσα ένα ερώτημα για το πότε θα κοιτάξουμε συνολικά το ζήτημα, όχι μόνο των σαρωτών, αλλά όλων ε, των συνδέσμων και με τις υπηρεσίες ασφαλείας ε, για να, να μπορέσουμε να το δούμε κάπως αυτό. Δεν αντιδράσατε σε αυτό από ό,τι κατάλαβα και αυτό και εγώ θα γίνει μέσω της τη επιτροπολογίας, αλλά μπορεί να απαντήσει ο κύριο Ρόιτε. Κύριε Γκράντε, θέλατε να πείτε κάτι? Ναι. Για τον τύπο, για την έκθεση έκανα μια έκθεση, αλλά με ανησυχεί και με ανησυχεί τι έγινε ακριβώς, ε, τι χρόνο διαθέτει για να την πρόθεση αυτής της ε, συζήτησης. Ε, έχει το χρόνο, διαθέτει χρόνο για να παρουσιάσει κανένα από τα βασικά σημεία. Σας ευχαριστούμε κύριε Ρόιτε, ένα λεπτάκι. Ναι, ναι, πάρτε το λόγο, αλλά ένα λεπτό μόνο. Όχι, εγώ ήθελα να ρωτήσω. Διαβουλεύτηκε η Επιτροπή με τον επιθεωρητή τον Ευρωπαίος για τη λύση αυτή με τον αρμόδιο. Ακριβώ αυτή ήταν η ερώτησή μου. Πολύ ωραία. Κύριε Ρόιτε, πείτε μας ακριβώς ποια είναι η διαδικασία και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα γιατί αυτό έχει προκαλέσει σύγχυση από ό,τι φαίνεται. Συγγνώμη δεν απάντησα στο ερώτημα αυτό. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι ε, ήρθαμε σε επαφή με τον ε, υπεύθυνο για την προστασία των ε, προσωπικών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προτού προχωρήσουμε με οποιαδήποτε επιπλέον νομοθεσία θα πρέπει να εξασφαλίσουμε προφανώς ότι έχουμε και τη δική του σύμφωνη γνώμη. Όσον αφορά το τι θα κάνουμε, τα πράγματα είναι σαφή. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι θα πρέπει να τροποποιήσουμε το παράγωγο δίκαιο, επομένως χρησιμοποιούμε τη δικασία της επιτροπολογίας και αυτό θα γίνει σε δύο επίπεδα. Το πρώτο, διαδικασία επιτροπολογίας που θα μας επιτρέψει, που θα σας επιτρέψει να έχετε το δικαίωμα κυρίας, δηλαδή να μην προσταθούν στον κατάλογο σαρωτές σώματος και στη συνέχεια θα έχουμε την τροποποίηση των εφαρμοστικών κανόνων όπου θα προσπαθούμε να διευθετήσουμε όλα τα ζητήματα προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχει κανένας κίνδυνος για την υγεία, θα προσπαθούμε να δούμε ποιο είδος μηχανισμού θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και γενικά θα προσπαθήσουμε να αφαιρθούμε σε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει ως ανησυχίες, προκειμένου να συμμορφώνεται κάθε κράτος μέλος με τους κανονισμούς αυτούς κάθε φορά που αποφασίζει να χρησιμοποιήσει τους αρωτές σώματος, είτε κατά αποκλειστικότητα σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους ελέγχου. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα. Είπαμε ότι θα κάνουμε μία αξιολόγηση αντικτύπου, η οποία θα ξεκινήσει ως Σονούπο. Και αυτό μπορώ να σας πω μια εκτίμηση κάνω. Μέχρι τα τέλη του έτους θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η αξιολόγηση, αυτή η μελέτη. Αυτή είναι η καλύτερη δυνατή εκτίμηση που μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή. Προφανώς όμως, στα πλαίσια αυτά η συζήτηση που θα γίνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η συζήτηση που θα γίνεται στο Συμβούλιο από τους Υπουργούς θα είναι πάρα πολύ σημαντική και για μας, προκειμένου να καταφέρουμε να δούμε πώς θα πρέπει να διαμορφωθούν και τι θα πρέπει να περιέχουν οι εφαρμοστικές διατάξεις και υπάρχουν κάποια σημαντικά ζητήματα, κάποια σημαντικά ερωτήματα. Τι είδους τεχνολογία θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Αν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι ακτίνες χ οπισθοσκέδασης. Επίσης, δεύτερον, τι είδους τεχνολογία θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να μην υπάρχουν προβλήματα υγείας κτλ. Και εκεί δίστανται λίγο οι απόψει μεταξύ ημών και ε, της κυρίας Λάτφορτ. Υπάρχουν διαφορετικά τύποι, διαφορετικοί τύποι μηχανημάτων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Θέλουμε λοιπόν ακριβώς να δούμε ποια είναι η τεχνολογία η οποία θα χρησιμοποιηθεί και πώς θα καταφέρουμε να έχουμε μία τεχνολογία η οποία θα συμμορφώνεται με όλες τις ανησυχίες που έχουμε εκφράσει και στο παρελθόν, ακόμα και πριν από δύο χρόνια, όταν λέγαμε ότι θα μπορούσαμε τότε να χρησιμοποιήσουμε χι αριθμό τεχνολογιών. Πρέπει λοιπόν να γίνει μία συζήτηση για τεχνολογία που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να μην υπάρχουν ανησυχίες ούτε για την προστασία των δεδομένων, ούτε για την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίασή σας, για τις απαντήσεις σε ερωτήσεις των βουλευτών. Και αναλόγως θα κινηθούμε και εμείς, είμαι σίγουρος. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Okay, next item on the agenda. Λοιπόν, επόμενο σημείο Συνημερίς για διάταξη. Έκθεση STEX διατυπώσεις ε, για τα πλοία. Έχουμε μείνει λίγο πίσω, με συγχωρείτε λοιπόν. Έχετε τον λόγο και παρακαλώ να αποχωρήσετε ε, ήσυχα και αν έχετε κάποια συνάντηση παρακαλώ εκτός έτους. Κύριε Στέρξη, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε και θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα όλους και μια συμφωνία με το Συμβούλιο που θα έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε μία μόνο ανάγνωση και να μπορέσουμε να εγκρίνουμε το κείμενο τώρα στην ε, Ολομέλεια του Ιουλίου. Και το κείμενο είναι στην, ατζέντα, στην ΟΕΣ διάταξη στις 23 Ιουλίου. Οπότε ας δούμε το τι έχουμε επιτύχει και το τι δεν έχουμε επιτύχει. Γιατί έχω την αίσθηση πως τη Δευτέρα ε, όταν επιτύχαμε συμφωνία πως ε, έκανα πολλές παραχωρήσεις. Και θα μπορούσαμε ίσως να επιτύχαμε ε, να έχουν επιτύχει πολύ περισσότερα πράγματα, αλλά αυτό το έχει κάνει πάντα στις διαπραγματεύσεις. Σε μπάση περιπτώσει, θεωρώ πως έχουμε επιτύχει την αρχή της απλοποίησης διαφόρων διατυπώσεων και ήταν κρίμα το ότι στη συζήτηση τα κράτη-μέλη κοιτούσαν μόνο το κόστος της υπόθεσης, το κόστος της οργάνωσης και όχι ποτέ το όφελος. Δηλαδή το πώς θα διευκολύνουμε και το εμπόριο και το πώς θα ωφεληθεί το περιβάλλον. Οπότε μιλάμε για μια εναρμόνιση των διατυπώσεων. Δεύτερον, η ηλεκτρονική ανταγραφή ανταλλαγή των δεδομένων, δηλαδή να μην χρειάζεται να δοθούν τα ίδια δεδομένα πολλές φορές, αλλά να περνάει ένα ηλεκτρονικό έντυπο σε ένα σύστημα και το σύστημα αυτό να φροντίζει να φτάνουν τα δεδομένα εκεί που πρέπει. Και σημαντικό είναι αυτό το οποίο ονομάσαμε στα αγγλικά single window ένα ενίο παράθυρο από το οποίο θα βγαίνει κανείς. Δηλαδή σημαντικό είναι οτιδήποτε αφορά την αυσιπλοεία και από το SafeSynet και ό,τι αφορά τα τελωνία και οτιδήποτε άλλο πιθανώς προσθεθεί μετανάστευση, λίστες επιβατών, πληρώματος όλα αυτά να ε, είναι διαθέσιμα σε ένα ενιαίο παράθυρο. Και πρόσθεσε το Κοινοβουλίο εδώ πέρα την εμπιστευτικότητα των δεδομένων και ε, έχουμε και απαλλαγή για πλοία που πάνε μεταξύ λιμένων Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία επί της αρχής δεν θα πρέπει να δηλώνονται. Βεβαίως, εντάξει, κάποιος κρατομέλος μπορεί για λόγους ασφάλειας ε, μετανάστευση να ζητάει δεδομένα, αλλά δεν θα είναι αυτός ο κανόνας. Αυτό το οποίο δεν μπορέσαμε να επιτύχουμε είναι πως ε, δεν θα είναι ένας κανονισμός με τη βάση φόρτωση πλοίων που πάνε σε τρίτη χώρα. Και εδώ πέρα ζητήσαμε από την Κομισιόν να το εξετάσει αυτό και να υποβάλει προτάσεις. Και μετά το έχουμε όλο αυτό σε ένα ξεχωριστό άρθρο, δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα τα οποία δεν έχουν λυθεί και αναμένουμε από την Κομισιόν να μας πει ποιε είναι οι δυνατότητες και τι μπορούμε να κάνουμε. Θεωρώ λοιπόν πως όταν μιλάμε για την αρχή της διοικητικής απλούστευσης των διαδικασιών θα επιτύχουμε αυτό το οποίο θέλουμε να επιτύχουμε δεύτερον υπήρχαν κάποια πράγματα τα οποία θέλαμε να προσθέσουμε. Πρώτα απ' όλα, μία γλώσσα. Αυτό δεν το συζητούσε το Συμβούλιο. Μας είχαν πει πως εάν χρησιμοποιήσουμε ε, τη λέξη γλώσσα είναι πρόβλημα και είναι πρόβλημα αυτό γιατί δεν γίνεται πολιτικά για το ε, Συμβούλιο και αν παραμέναμε στην αρχική τροπολογία δεν θα κινούνταν τίποτα. Οπότε βάλαμε κάποια πράγματα που λένε πως είναι σημαντική η γλώσσα. Αλλά υπάρχει μόνο ένα εκτιμώντας, δεν υπάρχει στα άρθρα. Και στο εκτιμώντας αυτό θα διαβάσω τώρα στα, στα αγγλικά γιατί με αγγλικά δουλέψαμε οι εθνικές απαιτήσεις γλώσσας συχνά είναι εμπόδιο στην ανάπτυξη των επάκτιων δικτύων αυσιπλοείας. Τα κράτη-μέλη πρέπει να καταβάλουν κάθε προσπάθεια να διευκολύνουν τη γραπτή και προφορική επικοινωνία μεταξύ κρατών μελών σύμφωνα με την διεθνή πρακτική με στόχο να βρεθούν κοινοί τρόποι επικοινωνίας. Όποιος το ερμηνεύσει αυτό βλέπει πως πρώτα απ' όλα είναι σημαντική η γλώσσα Δεύτερον, ζητάμε από τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε προσπάθεια έτσι ώστε γραπτός και προφορικά να διευκολυνθεί η επικοινωνία και τρίτον να έχουμε ένα κοινό μέσο επικοινωνίας. Εάν το μεταφράσουμε αν θέλετε αυτό, μιλάμε για τη χρήση μίας γλώσσας ή ενός συστήματος. και πηγαίνουμε προς τα εκεί που θέλουμε δηλαδή. Δεν χρησιμοποίησαμε τη λέξη γλώσσα και δεν λέμε ποια γλώσσα, αλλά μιλάμε για ένα κοινό μέσο επικοινωνίας γραπτής και προφορικής. Τι άλλο μπορεί να είναι αυτό πλην μιας γλώσσας. Τέλος πάντων. πετύχαμε κάτι το οποίο έστω δεν είναι στην αρχική μορφή. Δεύτερον, κάτι το οποίο ζήτησε το Κοινοβούλιο, για να δούμε τι θα γίνει με την εσωτερική ναυσιπλοεία. Ε, δεν είναι τόσο απλό αυτό τεχνικά. Αυτό το οποίο επιτύχαμε είναι να πούμε πως είναι σημαντική η εσωτερική πλοίο και έχουμε το άρθρο 11α στο οποίο ζητάμε ξανά από την Κομισιόν να μας δώσει αναφορά και να κάνει μία πρόταση. Να μας πει λοιπόν για δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα για το πώς θα επεκταθεί η απλοποίηση και δεύτερον το πώς θα ταιριάξουν μεταξύ τους ε, τα συστήματα τα θαλάσσια και τα ποτάμια. Οπότε νομίζω και εδώ πέρα βεβαίω δεν συμφωνούσε το Συμβούλιο, είπαμε πόσο σημαντικό είναι να πάμε όσο δυνατόν πιο πολύ μπορούμε ε, στην, στην ενδοχώρα, στην εσωτερική πλοία και να υπάρχει μια αρμονική λειτουργία. Τρίτον, που ήθελε να προσθέσει το Κοινοβούλιο, η σημασία των πλοηγών γιατί ε, λέγαν πως δεν υπάρχει κανένας λόγος να αφαιρθούν οι πλοηγοί εδώ πέρα. Εδώ πέρα μιλάμε για απλοποίηση διατυπώσεων και όχι για τους πλοηγούς. Αυτό το οποίο πετύχαμε τελικά είναι μια κοινή δήλωση Κομισιών και Συμβουλίου όπου λένε πως θα αναζητήσουν ένα ξεκάθαρο πλαίσιο για την απόδοση εξαιρέσεων στα πιστοποιητικά των πλοηγών. Οπότε βλέπετε στο 11α, να με συγχωρείτε, σε μια ξεχωριστή δήλωση, ζητάμε από την Κομισιόν πάλι να εξετάσει την όλη υπόθεση για να δημιουργήσει ένα σαφές πλαίσιο. Τα κράτη-μέλη θέλουν πρώτα ε, διαφορετικούς κανόνες ε, και να τους αναγνωρίσουν μετά αμοιβαία ενώ εμείς ζητάμε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Και αυτό το οποίο θεωρώ σημαντικό είναι πως μετά λέμε πως το πλαίσιο πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένο με αυτή την δήλωση, δηλαδή να, να έχουμε διοικητική απλοποίηση και με την ανακοίνωση της Κομισιόν για την Ευρωπαϊκή Λιμενική Πολιτική. Οπότε ε, έχουμε πει αρκετά πράγματα. Νομίζω πως με αυτά κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός και το ζήτημα των ε, πλοηγών έρχεται στο προσκήνιο και Συμβούλιο και Κομισιόν λένε πως θα το δούνε. Νομίζω και αυτή η δήλωση είναι θετική. Οπότε έχουμε τρία σημεία. Γλώσσα, εσωτερική νευσιβλοεία και πλοηγή που δεν τα ήθελαν και εμείς ε, καταφέραμε να βάλουμε μια δήλωση στην έκθεση ή ένα άρθρο στην οδηγία. ή ένα εκτιμώντας ή μια έκθεση της Κομισιόν ή μια δήλωση τέλο πάντων Συμβουλίου και Κομισιόν, κάτι επιτύχαμε. Ε, βεβαίως το δυσκολότερο ήταν η ημερομηνία. Πότε θα ξεκινήσουν όλα αυτά. Η Κομισιόν είναι Φεβρουάριο 2010, το Κοινοβούλιο ακολούθησε, η Κομισιόν μας έπεισε για κάποια πράγματα, μεταξύ των οποίων τα ηλεκτρονικά τελωνία και τα λοιπά. Ε, πώς ε, ήταν εφικτή η ημερομηνία. Δεν άκουγε τίποτα το Συμβούλιο, έλεγε πως έχουμε δυσκολίες, κόστος και είναι το 2017. Ε, Εμεί είπαμε πως είναι απαράδεκτο το 2017 και θέλαμε το 2013 και τελικά φτάσαμε στον Ιούνιο του 2015, δηλαδή το, τη μέση λύση αν θέλετε. Αυτό το οποίο επιτύχαμε είναι η προθεσμία για την εφαρμογή δεν θα είναι τα δύο χρόνια που προτείνει το Συμβούλιο αλλά 1,5 έτος κάτι μεταξύ δηλαδή αυτού πρότεινε Κομισιόν και Συμβούλιο. Σκέφτηκε πως εάν πρέπει να γίνουν αυτά στον ε, πραγματικό κόσμο και είμαστε έτοιμοι την 1η Ιουλίου 2014 να ε, μην έχουμε καμία διατύπωση στην ευσυπλογία τότε θα τα έχουμε πάει καλά και νομίζω αρχές 2013 είναι πάρα πολύ γρήγορα και υπήρχαν πάρα πολλές αμφιβολίες για το εάν θα είμαστε έτοιμοι. Και Εντάξει, μα είπαν ότι εσείς μπορεί να το θέλετε και να το κάνετε, αλλά ίσως δεν θα τα καταφέρουμε. Οπότε νομίζω πως ο Ιούνιος του 2015 είναι ένας καλός συμβιβασμό. Γιατί να ορίσουμε μια ημερομηνία έτσι ώστε τα κράτη-μέλη, τα λιμάνια να ξεκινήσουν να δουλεύουν. Αυτά επιτύχαμε να ευχαριστήσω τον συνάδελφο τον κύριο Μπεσέ που κατέθεσε τροπολογία για την ΕΜΣΑ την οποία απέσυρε γιατί η Κομισιόν είπε πως φέτος ήδη θα καταθέσει μία πρόταση για την ΕΜΣΑ και έχουμε τώρα στόχο να κατατεθεί όλο το κείμενο ως μία τροπολογία στην Ολομέλεια στην περίπτωση που θα έχουμε και άλλες τροπολογίες στην Ολομέλεια, το βεβαίω φεύγουμε από την συμφωνία. Νομίζω πως έχουμε μια τίμια ε, συμφωνία, ε, επιτύχαμε τους στόχους μας και έχουμε ένα σημαντικό βήμα για την εσωτερική αγορά όσον αφορά την ακτοπλοεία. Ζητώ λοιπόν από τους συναδέλφους να το σεβαστούν και να το υπερψηφίσουν την Ολομέλεια, στην Ολομέλεια τον Ιούλιο. Και να έχουμε έτσι μια ε, οδηγία η οποία θα τεθεί ενισχύ σε κάποια χρόνια και θα βοηθήσει και το εμπόριο και το περιβάλλον. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Στέρξ για την παρουσίαση που μας κάνατε. Ο κύριος Δεγκράντες Πασκουάλ για το ΕΛΚ. Sí, gracias, señor presidente. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Στέρκα, ε, μέσω της ευγένεια είμαι υποχρεωμένος ε, ε, να σας συγχαρώ πάντως. Ε, επειδή είστε και ευγενικός να συγχαρώ για την πολύ καλή διαχείριση όλων αυτών των θεμάτων. Νομίζω ότι οδηγείτε στο σωστό λιμάνι αυτή την πρωτοβουλία. Τώρα, πέρα μετά από τη συζήτηση και τα συμπεράσματα εδώ της Επιτροπής, έγινε μία ανάλυση ότι δεν θα υπήρχαν κανονικά ιδιαίτερες διαφορές. Και η κατάληξή μας ήταν ότι θα έπρεπε να δώσουμε μία εντολή στον εισηγητή για να διαπραγματευτεί έτσι ε, με το Συμβούλιο όπως πρέπει και να πετύχουμε τους δυνατούς στόχους το καλύτερο είναι ο εχθρό του καλού, λέμε πολλές φορές, αλλά νομίζω ότι με αξιοπρέπεια έκανε τη δουλειά που έπρεπε χωρίς να απαρνηθεί τις αξίες μας εδώ στην Επιτροπή και τον έκανε με επιτυχία. Σύμφωνο ιδιαίτερα λοιπόν από πλευράς της ομάδας μου του ΕΛΚ ε, να τεθεί έτσι με αυτούς τους όρους και θα δούμε και για τις τροπολογίες τον Ιούλιο και θα δούμε ίσως μια ενιαία ανάγνωση, μια και μόνο ανάγνωση. Τώρα τα προβλήματα είχαν να κάνουν με αυτά που είπε, όπως είπε το γλωσσικό από την άλλη μεριά. Τι έγινε τώρα, πώς θα καταλάβει ο Βέλγος τα προβλήματα τα γλωσσικά, λέγαμε στην αρχή, όμως ε, καταλάβαμε στον άλλο. Και στην περίπτωση αυτή, στα πλαίσια, μια ρύθμιση στα πλαίσια του, της έκθεσης ε, δεν ήταν πρόβλημα της ε, ε Ισπανικής Προεδρίας ε, ήταν η άρνηση διαφόρων χωρών που είχαν πολιτικό βάρος, συμβαίνει αυτό πολλές φορές και έχουμε μια κατάσταση που τον έχει κανείς δίκαιο τον κάνει να προχωράει όπως πρέπει και είναι προσπάθεια λοιπόν εξαίρεση λύσης ε, στην ελληνική έκθεση όχι τώρα ε, κάτι το σκέτο έτσι γιατί νομίζω ότι θα μπορούσαμε να δούμε και στο μέλλον για το ναυτικό δίκαιο της εκφράσεις όπως ε, θα πρέπει. Τώρα κάτι ακόμα ήταν μια ενιαία μορφή, ήταν δύσκολο όλα αυτά να λυθούν αποτελεσματικό. Αυτό για την ε, προθεσμία, για τη θέση σε ισχύ για όλους τους σοβαρούς ε, συζητητές όπως τον κύριο Στέρκ είναι κάτι που επαναλαμβάνεται εδώ η Επιτροπή λέει κάτι ναι εντάξει το αισιόδοξο για μια διαπραγμάτευση κάπου εδώ κοντά το Συμβούλιο η τάση του είναι να καθυστερήσει κάπως και η Επιτροπή μας θέλει να είναι ο εξορροπητικός παράγοντας. Νομίζω ότι η προθεσμία σας είναι λογική και ικανοποιεί τους πάντες. Τώρα, το να πετυχαίνουμε μια λύση είναι κάτι το θετικό σε αυτήν την υπόθεση και το κάνουμε έτσι χωρίς να καθυστερούμε τρομερά είναι καλό, γίνεται όπως είδαμε. Να μην ξεχνάμε κάτι ότι πρόκειται για ε, κάτι που έχει ένα πλαίσιο στα πλαίσια μιας ε, ε, μεταφοράς ε, ναυτιλιακής χωρίς ε, σύνορα, χωρίς εμπόδια μάλλον. Και με τον τρόπο αυτό θα βοηθήσουμε για όλες αυτές και τις συνδυασμένες μεταφορές και μάλιστα θα μειώσουμε τις διατυπώσεις που χρειαζόταν και που καθιστούσαν αργή τη μεταφορά και δύσκολη κάτι που στα πλαίσια αυτής της συνδυασμένης μεταφοράς έχει μεγάλη σημασία. Τώρα Εάν δεν είμαστε υπέρ της αποτελεσματικής δυνατότητας των υπολείπων και ευνοούμε μόνο μία, τότε πώς θα πετύχουμε αυτή τη συνδυασμένη μεταφορά, απλά και μόνο θεωρητικά ρητορικά θα το εξετάζουμε και τίποτα άλλο. Εμείς και από το ΕΛΚ είμαστε υπέρ με την ε, άποψη του κύριου Στέρκ. Ε, νομίζω ότι έκανε το έργο του όπως έπρεπε και σύμφωνα με τον Λέλη που του δόθηκε και θα μπορούσε να φτάσει στην Ολομέλεια ε, με μια συγκεκριμένη θέση για τα πάντα. Εντάξει, ίσως κάποιος να βρει κάποιο σημειάκι που να μην το αρέσει. Πάντως το σύνολο είναι καλό και θα ήθελα να συγχαρώ και πάλι τον κύριο Στέρκ. Κύριος ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος. Σε συνεννόηση με τον σχεδόν Συγκητή τον Κούντο Μιλάνα που απουσιάζει, θέλω να πω πως εμείς ως Σοσιαλδημοκράτε σας στηρίζουμε. Συμφωνούμε να κατατεθεί αυτό ως μία τροπολογία και να μην καταθέσουμε καμία άλλη τροπολογία. Νομίζω πως το πακέτο είναι καλό, και υπό λοιπόν την έννοια ότι θα οδηγήσει σε διοικητική απλούστευση ειδικά όσον αφορά την ενδοευρωπαϊκή ακτοπλοεία και θα οδηγήσει σε λίγο περισσότερη ανταγωνιστικότητα στον τομέα αυτών σε σχέση με άλλους τρόπους μεταφοράς ε, που λειτουργούν μια χαρά χωρίς πάρα πολλά χαρτιά στην εσωτερική αγορά Οπότε είναι ένα συν και σημαντική πρόοδος. Τώρα, οι διάφοροι συμβιβασμοί με το Συμβούλιο, νομίζω πως οι περισσότερες περιπτώσεις είναι επιτυχής, ειδικά όσον αφορά τους πλοηγούς. Αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο λέτε, πως η Κομισιόν θα πρέπει να κάνει μια πρόταση, δεσμεύεται να κάνει μια πρόταση Νομίζω πως θα είναι κάτι θετικό αυτό. Όσον αφορά τη γλώσσα, ναι, υπάρχει μια κατεύθυνση που δεν είναι βέβαια τελείω συγκεκριμένη. Αλλά νομίζω πως είναι πολύ ευαίσθητο να πάμε πολύ παραπέρα. Και θα πρέπει να δούμε και ποιες είναι οι ημερομηνίε έναρξης του κανονισμού δεδομένου των όσων είπατε για το ζήτημα των παρατηρήσεων αυτών θα μπορούσε να ξεκινήσει ένα χρόνο νωρίτερα δεν νομίζω να έχουμε κάποια προβλήματα συνοψίζοντας λοιπόν υποστηρίζουμε την πρότασή σας και θα την εγκρίνουμε unblock ευχαριστώ η πράσινη. Ο κύριος Μπεσέ. Γρήγορα και πολύ γρήγορα μάλιστα να κάνω μερικές παρατηρήσεις, ε, δηλαδή υπέρ των όσων λέει ο κύριο Τέρκ και χάρη στην εργασία του πετύχαμε μια ισορροπημένη θέση, ιδιαίτερα θετική σίγουρη, σίγουρα παρά το στη δύσκολη θέση από πλευράς ε, του Συμβουλίου όσον αφορά το χρόνο, τα μέτρα κλπ. Η εντύπωσή μας ήταν ότι είχαν ε, σηκώσει το χειρόφρενο σε κάθε φάση, σε κάθε στάδιο. Ο στόχος φαίνεται καθαρά, εκφράζεται καθαρά, σε εμά είναι ιδιαίτερα αξιόλογος και για μας τους οικολόγους, τους πράσινους και με ιδιαίτερη διάθεση να ευνοήσουμε την θαλάσσιες μεταφορές σε σχέση με άλλες μεταφορές που καταστρέφουν πολύ περισσότερο και την οικονομική μας ισορροπία και την οικολογική ισορροπία του πλανήτη μας. Εντάξει, σίγουρα γίνονται βήματα προς τα εμπρός, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά τα παρήθμισε ο κύριος Τέρκ και γίνεται ιδιαίτερα δεκτή η συμβαστική λύση, την αποδεχόμαστε. Τώρα το εμπόδιο δεχόμενο θα μπορούσε να είναι η ημερομηνία. Αποκλείεται, αποκλείεται να καθυστερήσουμε ακόμα το 1η Ιουλίου Ιουνίου του 2015 που είχε χανορίσει όλοι που συμμετείχαν στην εργασία του κυρίου Στέρκ. Αυτά λοιπόν δεν θα πρέπει να την ξεπεράσουμε την ημερομηνία. Λυπάμαι που η κοινή γλώσσα είναι κάτι το που προβάλλεται δειλά και θολά. Θα ήθελα περισσότερη έτσι βεβαιότητα, δεν θα ασχοληθώ όμως με λεπτομέριούλες. Είναι καλή αυτή η δουλειά και ε, η ομάδα μου ακριβώς η πράσινη θα είναι υπέρ αυτή της έκθεσης του κυρίου Στέρκ. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα Χαίρομαι για τους επένους που ακούγονται για τον κύριο Στέρξη γιατί δούλεψε σκληρά. Να ξεκινήσω από το τέλος. Το 2015 είναι αργά. Αν θέλουμε να επιτύχουμε κάποια βελτίωση. Μια εφαρμογή της σημερινής τεχνολογίας και απλοποίηση της γραφειοκρατίας και να περιμένουμε τόσο, τέλος πάντων. Τώρα για την ηλεκτρονική τεχνολογία και το ενιαίο παράθυρο είναι κάτι το πολύ θετικό και η προστασία των δεδομένων και νομίζω για τα πράγματα τα οποία δεν επιτύχαμε είναι κρίμα το ότι δεν τα επιτύχαμε αλλά υπάρχουν νομίζω προοπτικές ε, όσον αφορά και την γλώσσα σωστά το είπε ο κ. Στέξα έπρεπε να έχουμε τα αγγλικά όπως είναι και στην αεροπορία και αυξήθηκε η ασφάλεια και θα είναι και λογικό πρέπει να επιμείνουμε και να δούμε τι θα γίνει. Όπως και στην εσωτερική ναυσιπλογία που θα πρέπει να συμπεριληφθεί. Δεν ξέρω γιατί δεν το θέλουν τα κράτη μου Απορώ γιατί είναι πεπισμένη για τη σημασία της και για τους πλοηγούς. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον και να επιμείνουμε. Και νομίζω θα καταφέρουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Φαντάλεν τελικά. Ναι, κύριε Πρόεδρε, ο στόχος νομίζω επετεύχθη και αυτό μετράει. Θα γίνει καψιόπλωστερη ναυσιπλοεία και η ακτοπλοεία μεταξύ λιμένων της Ένωσης και θα έχουμε ένα βήμα προς τα μπρος για την εσωτερική αγορά και αυτό μετράει. Γι' αυτό και εγώ και η ομάδα μου θα υποστηρίξουμε την μία και μόνη σας τροπολογία. Η ημερομηνία δεν ξέρω αν είναι τόσο ρεαλιστική. Ίσως ε, βλέπω εκεί πέρα έχουμε άλλες συζητήσεις κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω. Ε, είναι ρεαλιστική η ημερομηνία γιατί πρέπει να υπάρξει πολλή εργασία για να καταλήξουμε σε κάποια αποτελέσματα. Οπότε εγώ δεν έχω πρόβλημα με την ημερομηνία εντάξει, τώρα για τη γλώσσα, αν άκουσα καλά, υπάρχει μία σαφής διατύπωση και μπορούν τα κράτη-μέλη να αποφασίσουν το τι θα κάνουν και ξέρουμε βεβαίω τι θα γίνει. άκουσα στην περίπτωση στην οποία η Κομισιόν ε, το θεωρήσει απαραίτητο θα καταθέσει πρόταση. Αυτό είπε ο κύριος Στέρξ. Υποθέτω πως η Κομισιόν θα μας πει πως εάν δεν θεωρεί απαραίτητη μια πρόταση να μας πει και το γιατί, ε. Ή θα ήθελα να μας το διευκρινίσει αυτό ο κύριος Στέρξ. Και τέλος, για τους πλεγούς, πράγματι καλό είναι να έχουμε ένα σαφές πλαίσιο. Από τα τρία σημεία αυτό είναι το καλύτερο. Οπότε θα ήθελα και μια διευκρίνηση ώστε να την στην κοινή ευλογία, κύριε Στέρξ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την Κομισιόν και ο, ε, κυρία, ο κύριος Θεολογίτης. Αν δεν υποστώ το όνομά σας, με συγχωρείτε. Thank you very much, Mr. Chairman, for giving... Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Θεολογίτης ονομάζομαι και εκπροσωπώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει. Θεωρώ μάλιστα ότι είναι ιδιαίτερα μετροπαθής όταν αναφέρθηκε στα όσα έχει επιτύχει, γιατί στην ουσία, αν μου το επιτρέπετε, έχει καταφέρει να επανεκαθιδρύσει κάποια από τα σημεία που ενδεχομένως να χάναμε από την πρόταση, αν οι συνάδελφοι από το Συμβούλιο τελικά περνούσαν την δική τους την τοποθέτηση. Και νομίζω το πιο σημαντικό σημείο που κατάφερε να περισσώσει είναι το single window, αυτό το ενιαίο παράθυρο. Χάρη λοιπόν στον εισηγητή, καταφέραμε να προωθήσουμε και το σύνολο της ε, ανακοίνωσης ε, αυτής και τα επιμέρους σημεία. Θέλουμε να έχουμε ένα σύστημα το οποίο δεν θα περιλαμβάνει κανένα εμπόδιο όσον αφορά τις μεταφορές και για να χρησιμοποιήσω και τα λόγια του Αντιπροέδρου και Επιτρόπου για τις μεταφορές του κυρίου Κάλλας, πραγματικά πρέπει να διατηρήσουμε τις προσπάθειές μας στον τομέα της καινοτομία και της τεχνολογίας, προκειμένου να διευκολύνουμε την εργασία των πολιτών μας και την ε, ζωή των ε, διοικητικών υπηρεσιών. για τα επιμέρους σημεία τα οποία στήξατε και για τα οποία εμείς πρέπει να υποβάλουμε μια έκθεση. Τα λαμβάνουμε λοιπόν υπόψη μας, όλα έχουν καταγραφεί σωστά και τα πάντα λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Και εμάς μας απασχολούν τα σημεία αυτά στα οποία αναφέρθηκαν οι ευρωβουλευτές και θα αναφερθώ σε ορισμένα από αυτά. Η ενσωμάτωση της ε, εσωτερικής ναυσιπλοείας και των εσωτερικών θαλάσσιων ποτάμιων οδών στην γενικότερη στρατηγική που έχουμε για τις θαλάσσιες μεταφορές. Του χρόνου ελπίζουμε ότι θα υποβάλουμε μία πρόταση για το e-maritime, τις ηλεκτρονικές θαλάσσιες μεταφορές. Θα συνεχίσουμε κατά αυτόν τον τρόπο τα όσα έχουμε ήδη ξεκινήσει με την πρόταση αυτή και θα καταφέρουμε επίσης να βελτιώσουμε και άλλες νομοθεσίες του παρελθόντος όπως αυτή που δημιούργησε το SAFE Sinet. Στη συνέχεια θα έχουμε την οδηγία αυτή για τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία και στη συνέχεια θα έχουμε μία άλλη νομοθετική πράξη που θα έχει να κάνει με τις ηλεκτρονικές θαλάσσιες μεταφορές με το e-maritime. Βλέπετε λοιπόν ότι η ε, Όλη η προσπάθεια πρόκειται να συνεχιστεί και στο μέλλον, σε καμία περίπτωση δεν σταματάει με την πρόταση αυτή και ε, στηριζόμαστε και στην υποστήριξη λοιπόν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ε, χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε την υποστήριξη των σχεδόν εισηγητών και όλων των πολιτικών ομάδων. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, και για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να μειωθεί το διοικητικό άχθος στο συντομότερο δυνατό και γι' αυτό το λόγο αναφερόμαστε στην αυτόματη ανανέωση που θα γίνει μέσω των πράξεων κατά εξουσιοδότηση και στην Κορεπέρ μεθαύριο νομίζω ότι θα κυριαρχήσει τελικά η λογική και θα καταφέρουμε να εγκρίνουμε και το σύστημα των πράξεων καταξιοδότηση και για αυτόν τον τομέα τον οποίο συζητάμε. Νομίζω ότι θα είναι προς όφελος όλων. Σας ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Για τις πράξεις κατά ακολουθούμε την γενικότερη προσέγγιση που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και που εξέφρασε και μέσα, μέσω μιας συγκεκριμένης έκθεσης για το ζήτημα αυτό. Δεν ξέρω αν ο Στέρεξ θέλει να προσθέσει κάτι ακόμα. Όχι. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους ε, που συνεργάστηκαν και τους συνεργάτες των συναδέλφων. Και νομίζω πως θα έχουμε πλειοψηφία για το κείμενο. Το κείμενο δεν το έχουμε εδώ και πολύ καιρό. Ε, ούτως ή άλλως το έχουν σκιώδεις ε, εισηγητές, οπότε είναι στην διάθεσή σας για να απαντήσω το ερώτημα του κυρίου Φαντάλν για την εσωτερική ναυσιπλοεία υπήρχαν κάποια προβλήματα που δεν μπορούσαμε να λύσουμε, γιατί είχαμε πρακτικές δυσκολίες, παραδείγματο χάρη το πρόβλημα αυτό με την εσωτερική ναυσιπλοεία. Γι' αυτό στο 11α είπαμε πως η Κομισιόν πρέπει να κάνει μια έκθεση. Σε διάστημα τριών ετών. Έχουμε δηλαδή 1,5 έτος ε, και άλλο ένα 1,5 έτος εντός του οποίου θα διερευνηθεί η δυνατότητα απλούστευσης και για την ιστορική νοσηλεία. Αν μπορεί ή όχι, γιατί δεν είναι τόσο απλό. Δεύτερον, οι υπηρεσίες πληροφόρησης υποτάμιας, εάν είναι συμβατές με αυτά τα οποία προβλέπονται στην οδηγία και με αυτά τα οποία υπάρχουν και τρίτον, πώς θα προχωρήσουμε περαιτέρω όσον αφορά το συντονισμό και την εναρμόνιση. Τέταρτον, εάν είναι δυνατόν, εάν μπορούμε, για πλοία τα οποία έχουν πάει σε τρίτη χώρα να προσαρμοστεί και εκεί πέρα η απλοποίηση. Γιατί υπάρχουν δυσκολίες με τα τελωνία και πρέπει να διερευνήσουμε το πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Και πέμπτο, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν έχουμε τόσα πολλά δεδομένα για το πόσα πλοία πλέουν εντός της Ένωσης και πόσα πλοία προέρχονται από τη Ρωσία ή στη Βόρεια Θάλασσα ή από την Αλγερία, από το Μαρόκο. Όλα αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά για να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Για όλα αυτά λοιπόν θα κάνει μια έκθεση Κομισιόν και εάν χρειάζεται, αλλά αυτό πάντα έτσι το λέμε και μπορούμε πάντα ούτως ή άλλως φιλικά να πούμε στην Κομισιόν πως θέλουμε να, να κάνει κάτι γιατί έχει ούτως ή άλλως το, το μονοπόλιο για αυτά τα πράγματα. Εάν λοιπόν το θεωρηστώ θα καταθέσει μια νομοθετική πρόταση. Για να δούμε λοιπόν σε ποια κατεύθυνση θέλουμε να πάμε. Και εδώ πέρα με αυτό συμφωνεί και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Γιατί δεν ήθελε να πει τίποτα το Συμβούλιο, οπότε απευθυνόμαστε τώρα προς την Κομισιόν να διαρευνήσει και πιθανώς, εάν χρειάζεται δηλαδή, να δούμε τι θα κάνουμε. Οπότε για να ενθαρρύνουμε την ακτοπλοεία και να έχουμε έναν ενιαίο χώρο, γι' αυτό ακριβώς υπάρχει αυτό το ρητό αίτημα Συμβουλίου και Κοινοβουλίου να το, κάνει, να το διερευνήσει η Κομισιόν. Και πρέπει να πω πως εγώ Εντάξει, δεν το ομολογώ, δεν το έχω αντιληφθεί πλήρω το, το ζήτημα. Το οποίο, για το οποίο αναμένω βεβαίω την ε, άποψη τη νομική μας υπηρεσία και βεβαίω αναμένω και το τι θα προκύψει και από την ε, Κορεπέρ. ευχαριστώ του συναδέλφους. Ε, Σας ευχαριστούμε κύριε Στέρξ. Να πω κι εγώ κάτι. Να πώς θα πρέπει να γίνονται τα πράγματα Δεν θα ήθελα να πάμε στην κατάσταση άλλων επιτροπών. Πάντως, όταν έχουμε εισηγητέ που κινούνται μόνοι τους τελικά, ατομικιστικά και δεν αντικατοπτρίζουν τη γνώμη της Επιτροπής, τότε συναντάμε μόνο προβλήματα και είχαμε το πρόβλημα αυτό την προηγούμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια. Στη συγκεκριμένη όμω περίπτωση, ο κύριο Στέρεξ εργάστηκε πάρα πολύ καλά με του και εισηγητέ, γνωρίζει πάρα πολύ καλά ποιοι είναι εντολή που του δόθηκε από την Επιτροπή μα επικοινώνησε πάρα πολύ καλά με τους υπόλοιπους συναδέλφους, συνεργάστηκε πάρα πολύ καλά με τους και ηγητές. Επομένω, Ντέρεξ, ευχαριστώ πολύ που εργάστηκες όπως έπρεπε να εργαστείς. Δεν είχα καμία αφιβολία, βέβαια ότι θα εργαζόσουν καλά. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια του Ιουλίου, έτσι δεν είναι, ναι. Η συζήτηση θα γίνει τη Δευτέρα το βράδυ και η ψηφοφορία φαντάζομαι ότι θα γίνει την Τρίτη. Ελπίζω, λέει ο Πρόεδρος. Όπως ε, γνωρίζεις, υπήρξε ανταλλαγή επιστολών μεταξύ ε, ε, μου και του Προέδρου του Κοινοβουλίου και ήθελα να το ρωτήσω αν τελικά πιστεύω ότι εμείς είμαστε η μόνη επιτροπή που επιθυμεί να ξενυχτά διαρκώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό το λόγο μας μετέφεραν από, το, από τα μεσάνυχτα σε απογευματινή συνεδρίαση. καταφέρουμε κατά αυτόν τον τρόπο να αποφύγουμε αυτές τις πολύ προχωρημένες βραδινές ώρες που μας έδινε αρχικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η συζήτηση λοιπόν θα γίνει την Δευτέρα και θα ψηφίσουμε την Τρίτη το μεσημέρι. Αυτά για την Ολομέλεια του Ιουλίου. Λύεται σε αυτό το στάδιο συνεδρίαση. Θα συνεδριάσουμε πάλι αύριο στι 9 το πρωί. Θα γίνει εκεί η ψηφοφορία. Ο πρόεδρο ευχαριστεί και του Δερμηνεί, καθώ επίση και του Δερμηνεί στην νοηματική γλώσσα.